Państwa, możemy chyba, czy powinniśmy już rozpocząć, bo zbliża się prawie... Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε, πέρασε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Ελπίζω να μην σας τρομάζει αυτός ο όγκος εγγράφων που έχετε μπροστά σας. Ξέρετε ότι στο τέλος του σχολικού έτους, πριν από τις θερινές διακοπές, προσπαθούμε να κλείσουμε όσο δυνατόν περισσότερα σημεία, περισσότερα ζητήματα, προκειμένου να πάμε λίγο πιο χαλαροί στις θερινές διακοπές, έχοντας ε, ήσυχη τη συνείδησή μας. Ελπίζω όμως ότι δεν έχουν ξεκινήσει για ορισμένου ήδη από σήμερα διακοπές. Ελπίζω να έρθουν και περισσότεροι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της ημέρας σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή μας συνεδρίαση. Έχουμε πολλά σημεία στην σημερινή ημερήσια διάταξη, τα οποία πιστεύω όμως ότι χάρη στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε θα καταφέρουμε να καλύψουμε αποτελεσματικά και γρήγορα. Και επίσης έχει γίνει μια πολύ καλή προπαρασκευαστική εργασία από τη Γραμματεία. Όσον αφορά λοιπόν την ημερήσια διάταξη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Ξέρετε ότι μεταδίδεται μέσω του δικτύου συνεδρίασή μας. Ας περάσουμε στις ανακοινώσει του Προέδρου. Προφανώς έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες. Εξαιρούνται 5 γλώσσες, οι οποίες δεν καλύπτονται. Δεν έχουμε τον κύριο Γλέζο σήμερα στη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι ε, ο συνάδελφός μας ε, Γλέζος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, ήταν ε, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής μας από την ΚΟΕ, παρετήθηκε. Παρετήθηκε από το Κοινοβούλιο. Το ευχόμαστε λοιπόν καλή συνέχεια. Τον ευχαριστούμε πολύ για την ενεργή συμμετοχή του στην Επιτροπή μας, για το ότι συμμετείχε πάντα πολύ ενεργά. Θα μας λείψει σίγουρα πολύ και ελπίζουμε να έχουμε και στο μέλλον τόσο ενεργά και δραστήρια μέλη στην Επιτροπή Γεωργίας και ας λάβουμε υπόψη επίσης και την ηλικία του συναδέλφου. Αλλά και η κυρία Πόλσεν επίσης πρόκειται να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα την έχουμε όμως λίγο ακόμα μαζί μας θα συνεχίσει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις Επιτροπής μας και ασχολείται με δύο σημαντικά ζητήματα. Θα μας λείψει όμως και αυτή πολύ σίγουρα. Αλλά το Σεπτέμβριο θα την αποχαιρετήσουμε επίσημα. Τώρα, η Διεύθυνση Νομοθετικών Πράξεων και Δραστηριοτήτων μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε μια σειρά από διορθωτικά κείμενα τα οποία μας έχει προτείνει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέσσερις κανονισμούς της κοινή γεωργικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 231 του κανονισμού. Τα διορθωτικά αυτά κείμενα τα έχετε στο φάκελό σας και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διορθώσεις. Τις παρουσιάζω πολύ γρήγορα. Έχουμε καταρχάς τον κανονισμό 1308 του 2013 Όσον αφορά την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, θα πρέπει ο κανονισμός αυτός να διορθωθεί σε τρία σημεία, στο άρθρο 230 σημείο 1, σημεία C και E, καθώς επίσης και στο παράρτημα 2 και στο παράρτημα 7. Στα σημεία αυτά πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Όταν ενοποιήθηκε το κείμενο αυτό του κανονισμού, παραλήφθηκαν κάποιες προσθήκες όταν κάποιες συμπεφωνημένες αλλαγές της τέταρτης στήλη ενσωματώθηκαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια έχουμε τον κανονισμό 1305-2013 για την άπτυξη Πέθρου και εδώ πέρα έχουμε κάποια διορθωτικά κείμενα στο σημείο ε του άρθρου 59.4 καθώς επίσης και στο παράρτημα 6. Οι διορθώσεις αυτές περιλαμβάνονται στο κείμενο το οποίο έχετε στο φάκελό σας. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την δική μας την Επιτροπή και θα επιβεβαιωθούν στη συνέχεια από την Ολομέλεια. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα σα παρουσιάζω τώρα εδώ σήμερα. Αν μέχρι το τέλος των εργασιών μας σήμερα δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, σας προτείνω να εγκριθούν τα διαφορετικά αυτά κείμενα. Πρόκειται για τεχνικά, τυπικά ζητήματα, αλλά ξέρετε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, να εγκρίνουμε εμεί πρώτα αυτέ τι διορθώσει και στη συνέχεια η Ολομέλεια. Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 26η Μαου, τη 8η Ιουνίου, τη 16η και 17η Ιουνίου. Αν δεν έχουν υποβληθεί παρατηρήσει μέχρι το τέλο τη σημερινή συνεδρίαση, θεωρούνται ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο 4 παρουσίασε της έκθεση της αποστολής αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας, στη Διεθνή Έκθεση Έξπο του Μιλάνου. Αποστολή που χώρα από τις 17 ως 19 Ιουνίου. Η κυρία Αγγιλέρα Γκαρθία θα μας ενημερώσει για την αποστολή αυτή. Στο πρώτο τμήμα της επίσκεψης αυτής προείδρευα εγώ και στη συνέχεια η αντιπροεδρό μα, η κυρία Γκαρθία Αγκουλέρα, γιατί εγώ χρειάστηκε να αποχωρήσω λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Δεκάστρο για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε τελικά να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή. Συνεπώς, ενδεχομένως θα πρέπει, κύριε Δεκάστρο να επαναλάβουμε την επίσκεψη αυτή, καθότι εσείς δεν ήσασταν παρόν δυστυχώς. Ενδεχομένως να κάνω κι εγώ κάποιες προκατακτικές παρατηρήσεις όσον αφορά την αποστολή αυτή, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Αντιπρόεδρο Γκαρθία Γκουλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία να είμαι μέλος της αντιπροσωπείας μας ε, στο Μιλάνο. Όλα τα μπορείτε να τα διαβάσετε στο έγγραφο το οποίο παρουσίασε η Γραμματεία. Θέλω να συγχαρώ τη Γραμματεία πρώτα απ' όλα για την προσπάθεια και το έργο που έχει κάνει και πριν ε, την ε, αντιπροσωπεία και στη διάρκεια και γιατί ήταν ιδανική τοποθεσία που μείναμε και τα περίπτερα που επισκεφθήκαμε στο Μιλάνο, αλλά και η επόμενη μέρα που πήγαμε στην κοινοπαραξία Γκόργοντζόλα και στο Μουσείο Φρατέλη Μπράνκα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και επικαιρή επισκέψη. Είδαμε το μουσείο, γνωρίσαμε τις ιδιαιτερότητες και την ε, ονομασία προέλευσης Γκοργοντζόλα. Θέλω να συγχαρώ τη γραμματεία για τη δουλειά. Δεν μπορούσε να παραμείνει ο πρόεδρος. Μα έλειψε και ο συντονιστής μας, ο Πάολο. Επιτρέψτε μου να το πω. Μα έλειψε σε αυτή την επίσκεψη. Γιατί είναι η ψυχή, αν θέλετε. Είναι... Ε, αυτός που εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για την ΕΞΠΟ και δεν μπόρεσε να έρθει τελικά. Εκπροσωπήθηκαν πάντως σε όλες τις πολιτικές ομάδες, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Και πραγματικά ήταν καταπληκτική και πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη στα περίπτερα. Είδαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται. Και κράτησα την προσωπική μου εμπειρία βέβαια. Είδαμε ότι εκεί δεν είναι μόνο μια έκθεση καταπληκτική παγκοσμία έκθεση, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ εσωτερική δουλειά που γίνεται εκεί. Και σίγουρα θα πρέπει η Επιτροπή μας, Επιτροπή μας να παρακολουθήσει όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στην έξπο του Μιλάνου. Έχετε παραλαμβάνω στο έγγραφο όλες οι λεπτομέρειες για αυτήν την επίσκεψη, ολοκληρώνοντας, επαναλαμβάνω πρόεδρε, καταπληκτική δουλειά η γραμματεία και εκ μέρους των συναδέλφων που ήμασταν παρόντες ε, ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία, το λέω εξ όλων και προσωπικά να επαναλάβω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ΕΚΣΠ και επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το διατροφικό σύστημα και μας ενδιαφέρει και μας ενισχύει το να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική εμπειρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Όπως είπε η συνάδελφος, έχετε την έκθεση αυτή από τη γραμματεία, έχει διανεμηθεί σε όλους σας. Εγώ να κάνω δύο σύντομες ε, προσωπικές παρατηρήσεις και είναι καθαρά προσωπικές, το τονίζω αυτό. Η διεθνής αυτή έκθεση του Μιλάνου μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κάποιες νέες ε, προτάσεις ε, στον τομέα της γεωργίας και νομίζω ότι ήταν πάρα πολλοί και επισκέπτες, αυτό το είδαμε επί τόπου. Επίσης, καταφέραμε να δούμε διάφορα νέα αρχιτεκτονήματα, συνέβαλαν πάρα πολλοί διάφοροι αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες προκειμένου να προτείνουν κάτι εντελώς διαφορετικό και ενδιαφέρον και να προσελκύσουν πάρα πολλούς επισκέπτες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όλες οι παρουσιάσεις γίνανε με καθαρά ηλεκτρονικό τρόπο. Οι παρουσιάσει αυτές ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε. και σίγουρα προσέλκυσαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον ιδίω των νέων επισκεπτών. Θα θέλαμε λοιπόν από τον συνάδελφο Ντεκάστρο να αποτιμήσει και αυτός την διεθνή αυτή έκθεση του Μιλάνου, καθώς επίσης και την επίσκεψή μας στην έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αποτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την σημαντικότητα αυτή έκθεση σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Ξέρετε ότι η ΦΑΟ προφανώς έχει την έδρα της στη Ρώμη και νομίζω ότι τέτοιες θετικές εμπειρίες θα μπορούσαμε να τα επαναλάβουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε και κάποια σημαντικά μηνύματα και διδάγματα τα οποία θα πρέπει να μας εμπνεύσουν και για άλλες τέτοιες θετικές εμπειρίες στο μέλλον. Αυτά είχα να πω εγώ. Να περάσουμε δεχομένως στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Έχουν φτάσει οι ομιλητές μας. Ο κύριος Δαντάν έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και με, εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτής της ε, έκθεσης. Και όπως είπε και η Αντιπρόεδρος, κυρία Αγγιλέρα, ε, θα περάσω και για τις διακοπές μου, κάποιες, στις διακοπές μου κάποιες μέρες αυτόν τον, προορισμό. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα είδαμε. Αλλά να πω κάποια πράγματα για το ευρωπαϊκό περίπτερο, το περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ειλικρινά, πάνω από 50 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιφορτισμένη με την δημιουργία της ευρωπαϊκής ε, γεωργικής πολιτικής και ευρωπαϊκής πολιτικής τροφίμων το θέμα της ΕΞΠΟ ήταν πάρα πολύ σημαντικό ε, για ένα με πολύ μεγάλο μέρος της κοινή γνώμης. Το περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν ήταν στο ύψος των προκλήσεων, για να μην πω ήταν εκτός θέματος. Ε, δηλαδή με χειμωριστικά σκίτσα μας δείχνει να συναντιέται ένας αστός με μια επαρχιοπούλα ή το αντίθετο κάτι τέτοιο. Ε, το λέω αυτό γιατί πραγματικά με απογοήτευσε το περίπτερο αυτό, το δικό μας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια ότι περί γράφεται ως ε, μία έκθεση που μπορεί να προωθήσει τις ε, βέλτιστες πρακτικές ε, για να σεβαστεί το έδαφος, παραδόσεις, το περιβάλλον, αλλά τελικά μεγάλη αντίφαση όταν δούμε ποια είναι η γεωργική πολιτική για τις ελεύθερες συναλλαγές, εκβιομηχάνηση της γεωργίας. Δεν ξέρω, όλα αυτά μου φαίνονται αντιφατικά. Bardzo dziękuję. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, όπως σας είπα θα μας δοθούν και στο μέλλον ευκαιρίες για να συζητήσουμε την έκθεση αυτή στο Μιλάνο και να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Πάντως σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και μπορούμε έτσι να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Przechodzimy do punktu piątego. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 5 της μερίσιας διάταξης. Εδώ έχουμε την παρουσίαση δύο ειδικών εκθέσεων που θα μας παρουσιάσει η κυρία Κέρστη Καλιούλαιτε η οποία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται λοιπόν για δύο εκθέσεις. Η πρώτη είναι η έκθεση υπαριθμών 4 του 2015 με τίτλο «Τεχνική συνδρομή» Ποια είναι η συμβολή της στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Η δεύτερη έκθεση, η υπαριθμών 5 του 2015, τυπλοφορείται «Είναι τα χρηματοδοτικά μέσα επιτυχημένο και πολλά υποσχόμενο εργαλείο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης». Θα θυμάστε ότι είχαμε μια παρουσίαση από τον αρμόδιο επίτροπο για τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Επομένω, οι δύο αυτέ εκθέσει είναι ιδιαίτερα επίκαιρε και θεωρώ ότι θα συμβάλλουν πάρα πολύ στη συζήτηση που θα κάνουμε. Στι 9 Μαρτίου, οι συντονιστέ τη Επιτροπή μα είχαν μια συνεδρίαση με μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου που ασχολούνται με αγροτικά ζητήματα μετά λοιπόν από την γόνιμη αυτή συζήτηση που είχαμε, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Και αποφασίσαμε επίσης να ενισχύσουμε και την ανταλλαγή πληροφοριών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα, στη σημερινή μερίσια διάταξη, έχουμε ενσωματώσει την παρουσίαση των δύο αυτών εκθέσεων. Η πρώτη έκθεση, όπως σας είπα, έχει να κάνει με την τεχνική συνδρομή είχαμε συζητήσει το ζήτημα αυτό και σε πρώτερη συνεδρίαση των συντονιστών, θεωρούμε ότι η τεχνική συνδρομή μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά στη διόρθωση του ποσοστού σφάλματος που παρατηρείται πολύ συχνά και μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική γεωργική πολιτική και πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Κάλιουλα, η οποία όπως σας είπα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα μας παρουσιάσει ίδια και τις δύο εκθέσει και στη συνέχεια, ο συνήθως, θα ακολουθήσει συζήτηση. Και θα ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας και στη συνέχεια θα μπορέσει να απαντήσει πάλι η κυρία Λάιντ. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ Νομίζω ότι όντως η συνδρομή που θα έχουμε με το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητική. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς μέλη της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Να προχωρήσω στην παρουσίαση και των δύο εκθέσεων. Εξαιρετική περίπτωση για μένα, διότι συχνά πηγαίνουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού γιατί οι εκθέσεις μας απευθύνονται στους νομοθέτες της ε, Επιτροπής εκείνης, αλλά και σε εσά. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει πολύ η συζήτηση μαζί σας. Πρόκειται για την ειδική έκθεση με τίτλο «Τεχνική συνδρομή. Ποια είναι η συμβολή της στη γεωργία και στην ε, αγροτική ανάπτυξη» για την διαχείριση της τεχνικής συνδρομής και της συμβολής της στις, ε, στους βασικούς στόχους της γεωργικής πολιτικής για τα έτη 2007 έως 2014. Οι ελεγκτές μας ε, εξέτασαν ποιες δραστηριότητες υποστηρίχτηκαν από τεχνική συμβολή στο επίπεδο της Κομισιόν και των χωρών μελών. Εάν τα κόστη που ε, επιλέχθηκαν, τα οποία ζητήθηκαν δηλαδή εκ των υστέρων από τις χώρες μέλη, είχαν, ήταν δικαιολογημένα. Η τεχνική συμβολή έχει σχέση με την παροχή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης της χώρες μέλη για την ανάπτυξη Και βεβαίω τα διοικητικά κόστη καλύπτονται, αλλά η χρηματοδότηση τη τεχνικής συμβολής θα πρέπει να συνεπιφέρει και πρόσθετη δημιουργία ικανοτήτων. Αυτό είναι και το βασικό κλασικό νόημα τη τεχνική συνδρομής. Οι χώρε μέλη είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση τεχνική συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για ορισμένε ευρέω ορισμένε δραστηριότητε μέχρι κατοφλίου μέχρι οροφής μάλλον 4% του σχετικού προϋπολογισμού. Για το 2007 2013 οι χώρες μέλη είχαν σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουν 1,5 δισεκατομμύριο. Για το 2014 μέχρι 20 το ποσό αυτό αυξάνεται το περίπου 1,9 δις δισεκατομμύρια ευρώ. Για να προσφέρει η προστιθέμενη αξία η τεχνική συνδρομή δεν επιτρέπεται να αντικαταστήσει την ε, τις διοικητικές δαπάνες, αλλά πρέπει να είναι χρηματοδότηση για καθημερινή χρήση για τα διάφορους σχεδιασμούς. Βέβαια, οι πόροι για τη χρησιμοποίηση, για την, για την οικοδόμηση ικανοτήτων έχουν χρησιμοποιηθεί και για να καλύψουν κενά σε διοικητικούς προϋπολογισμούς και για μισθούς σε, έναν, σε μια περίοδο που έχουν μειωθεί πολύ οι σχετικοί προϋπολογισμοί. Τέσσερις από τις, ελεγχόμενες, από τις πέντε ελεγχόμενες χώρες είπαν ότι τα διοικητικά έξοδα ήταν η μεγαλύτερη δαπάνη τους για, από την τεχνική συνδρομή. Από το 2007 έως 2013 τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν για επιχειρησιακές δραστηριότητες. Υπάρχουν όμως ορισμένοι δείκτες που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δα, ε, δαπανά έναν μέρος του προϋπολογισμού της για τεχνική συνδρομή και για διοικητικό κόστος, για την κάλυψη διοικητικού κόστους. Τώρα, η ανάπτυξη τεχνολογίας ε, ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων είναι δαπάνη τεχνικής συνδρομής, όχι όμως η συντήρηση των ε, ε, συστημάτων αυτών που είναι διοικητική δαπάνη. Και οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρήκαν οι ελεγκτές δαπανούν μέρος του προϋπολογισμού της τεχνικής συνδρομής για την κάλυψη διοικητικών δαπανών. Αυτό δεν το απαγορεύει βέβαια καταρχήν η νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι να ξοδεύονται χρήματα για μισθούς διοικητικών υπαλλήλων ή άλλα καθημερινά έξοδα δεν είναι η καλύτερη χρήση της χρηματοδότησης τεχνικής συνδρομής. Τα χρήματα αυτά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έργα ανάπτυξη της υπαίθρου επιτόπου Επομένω, είναι ευκαιριακό κόστο και καλύπτεται από τον ίδιο τον αγροτικό τομέα. Άρα τελικά καταλήγουμε σε λιγότερε πραγματικέ επενδύσει και περισσότερη διοίκηση. Η τεχνική συνδρομή δεν σημαίνει μόνο γεωργία και ανάπτυξη τη εμφανίζεται και σε άλλους τομείς της ε, χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω δεν είναι όλα άσχημα τα νέα δραστηριότητες Rural Networking επιτρέπουν την χρήση της τεχνικής συνδρομής μέσα στα πλαίσια του γεωργικού προϋπολογισμού. Αυτά τα ε, αγροτικά δίκτυα ή τα δίκτυα της υπέθρου που επιτρέπουν τη βελτίωση της συνεργασίας και την αύξηση της τεχνογνωσίας είναι κατάλληλο όχημα για την τεχνική συνδρομή. Τέλος, θέματα επιλεξιμότητας. Είδαμε μη ομαλές χρηματοδοτήσεις από τον πυλώνα της τεχνικής συνδρομής, αλλά τα βασικά προβλήματα για τη χρηματοδότηση των αστηριοτήτων και των δύο πυλώνων και επομένω δεν είναι επιλέξιμα πλήρω, αναφέρονται και σε ε, σύναψη συμβάσεων και στις προμήθειες. Μπορεί τελικά να προκύψει σύγχυση σχετικά με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ταμείων και για τη χρηματοδότηση υπό τον πυλώνα 1. Το γεγονός ότι το διοικητικό κόστος είναι επιλέξιμο για τον πυλώνα 2 μόνο ε, ή ότι η Κομισιόν θα πρέπει να τα διαιρεί ανάμεσα στους δύο πυλώνες σημαίνει ότι υπάρχουν περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες για να δικαιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε η κατανομή των δαπανών αυτών. Τώρα, στην αξιολόγηση το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε ότι ούτε η Κομισιόν ούτε οι χώρες μέλη έχουν θεσπίσει κατάλληλο πλαίσιο αποδοτικότητας για να καταδείξουν την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης τεχνικής συνδρομής. Να με επιτρέψετε τώρα να έρθω στα χρηματοδοτικά εργαλεία, αν επιθυμείτε. Αν θέλετε δηλαδή να αναφερθώ και στις δύο εκθέσεις. Α, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία μου. Ας ε, κάνουμε λοιπόν κοινή συζήτηση και των δύο εκθέσεων. Για τα χρηματοδοτικά τώρα ε, μέσα. Σε περίοδο σημαντικών περικοπών των δημοσίων προπολογισμών, για να γίνουν περισσότερε επενδύσει με λιγότερα χρήματα του δημοσίου, έχει μεγάλη σημασία. Αυτά τα financial instruments λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι σπάνιοι ε, κρατικοί πόροι μέσα στα πλαίσια του ίδιου προπολογισμού. Τα ταμεία αναμένεται να επαναχρησιμοποιήσουν τα αρχικά χρήματα και αυτό λέγεται revolving factor και να προωθήσουν περισσότερο την επιτευξιμότητα των στόχων με χρήση δημοσίου ή και ιδιωτικού κεφαλαίου. Και ιδιωτικού κεφαλαίου και αυτή, αυτό είναι το αποτέλεσμα της μόχλευσης. Οι χώρες μέλη έχουν ιδρύσει 11 ταμεία εγγύησεων και 3 ταμεία δανείων από το 2009 στο 2014, στα οποία τοποθετήθηκαν 700 εκατομμύρια ε, ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Για τη νέα περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί τον διπλασιασμό σε ορισμένους κέριους τομείς των επενδύσεων. Τρεις βασικές ερωτήσεις ίσχυαν για μας. Χρησιμοποιήθηκαν σωστά τα financial instruments το 2007-2013. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία απέδωσαν καλά στην περίοδο 2007-2013 και η περίοδος 14-20 προσφέρει την δυνατότητα των ε, αναγκαίων βελτιώσεων για το setup και την, ανακεφαλαιο... και την κεφαλαιοποίηση βρήκαμε ότι δεν είχε επαρκή βάση ε, τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία για, το 2000, για την περίοδο 2007-2013. Δεν υπήρχε πραγματική ζήτηση για χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα των γεωργικών επενδύσεων, όπως έδειξε η έρευνά μας για τις χώρες μέλη. Η ζήτηση στον τομέα της γεωργίας δεν είχε αξιολογηθεί σωστά και δεν είχαν ε, δοθεί επαρκείς ενδείξεις για τις ελλείψεις που διαπιστώνονταν στις χώρες μέλη. Οι κανόνες για την δαπάνηση έχουν οριπτώσει πλεονεκτήματα στις χώρες μέλη. Προκαταβολή των ε, δαπανών, συμβολές στα χρηματοδοτικά εργαλεία που ακόμα δεν έχουν όμως φτάσει μέχρι τους τελευταίους, ε, τελικούς μάλλον δικαιούχους. Οι εφαρμοστεί κανόνες επιτρέπουν τη δαπάνηση όλου, όλης της αξίας των εγγύσεων Σημαντικές λοιπόν ελλείψεις που οδήγησαν σε σημαντική υπερκεφαλαιοποίηση των ε, χρηματοδοτικών εργαλείων. Στην περίπτωση ιδέ των ταμείων εγγύσεων βρήκαμε ότι 421 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στο κεφάλαιο 11 ταμείων εγγύσεων όλες αυτές οι εγγυήσει, συνολικά δηλαδή περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσαν να είχαν, να είχαν βασιστεί σε ένα καταβληθέν κεφάλαιο της τάξης των 50 εκατομμύρων ευρώ. Υπήρξε λοιπόν μαζική υπερκεφαλαιοποίηση των ταμείων εγγυήσεων κατά τουλάχιστον 370 εκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, το ποσό αυτό είχε παγώσει χωρίς καμιά συμβολή σε εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών. Ακούμε συχνά ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να καταφέρουν περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα εδώ συνέβη το αντίστροφο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να προσφέρουν και τη δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων μέσω του, της, ε, της ε, διαδικασίας της μόχλευσης και του ε, revolving factor. Αυτό να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και ιδιωτικά κεφάλαια. Προσελκυστούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι ο revolving factor και το εφέ της μόχλευσης δεν ήταν επαρκή στην περίπτωση των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων για την περίοδο που έληξε το 2013. Οι χώρες μέλη δεν έπραξαν αρκετά για να επιτύχουν πραγματικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Δεν προσήλκησαν επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια για να εισρέψουν τα ε, ταμεία χρηματοδότησης για να οδηγήσουν σε ανάπτυξη στην, στον χώρο της υπέθρου. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν απέδωσαν το αναμενόμενο και δεν πρόσφεραν τα πλήρη ενδεχόμενα ε, θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την, ε, το αποτέλεσμα ανακύκλωσης και της μόχλευσης. Και αυτό είναι εν τέλει το ερώτημα. Επίσης, τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία ιδρύθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε τα χρήματα του δημοσίου να επιτρέψουν την προσέλκυση και τη χρήση και άλλων δημοσίων χρημάτων, επιδοτήσεων δηλαδή. Για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υλοποιήθηκαν το 2007-2013, το συνέδριο βρήκε ότι μόνο όσοι είχαν υποβάλει αιτήσει για επιδοτήσεις είχαν τελικά πρόσβαση σε αυτά. Δεν θα πρέπει όμω ο κοινοτικό προπολογισμό να είναι ο μόνο που αναλαμβάνει τον κίνδυνο για διάφορε επενδύσει. Όμω αυτό συνέβη τελικά. Τα συμπεράσματα των ε, ε, ελέγχων μα αναφέρονται στην εφαρμογή του, της περίοδου 2007 έως 2013. Πρέπει ωστόσο να εφαρμόσουμε τις αρχές στις οποίες έχουμε καταλήξει και για το 2014 έως 2020. Χρειαζόμαστε λοιπόν υποχρεωτικές εκ των προτέρων αξιολογήσεις για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, περισσότερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, οι βασικές μας ανησυχίες δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί, δηλαδή ο κίνδυνος υπερκεφαλαιοποίησης παραμένει. Οι δε όροι για την απόδοση δεν περιλαμβάνονται μέσα στους όρους χρηματοδότησης. Είναι θετική η πρωτοβολία του Επιτρόπου Χόγκαν για εντατικότερη χρήση των ε, χρηματοδοτικών εργαλείων στην επόμενη περίοδο. Επισημαίνω όμως ότι χρειάζονται όχι μόνο περισσότερα, και καλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης των ταμείων και ε, της ε, μόχλευσης χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση των δύο ειδικών εκθέσεων. Zgodnie i Σας ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν από λίγο, θα περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Γιάρ πρώτος, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μας επιτρέπει να διεξαγάγουμε τη σημερινή συζήτηση στην ουσία προβαίνεται σε αξιολόγηση ή κατά κάποιο τρόπο μας δίνεται και το πιστοποιητικό καλής διαγωγής. Εμείς κάνουμε την ομοθέσια, βεβαίως χρειαζόμαστε τον διάλογο μαζί σας για να δούμε αν πραγματικά τα νομοθετήματά μας αποδίδουν τα ποθούμενα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο που επιτρέπει τη συνέχεια αυτού του διαλόγου. Και ίσως μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποιους υπευθύνους οι οποίοι θα συνεχίσουν, να αναθέσουμε δηλαδή σε κάποιους, να συνεχίσουν τον διάλογο αυτό. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τις εκθέσεις, έτσι λοιπόν θα περιοριστώ μονάχα στα όσα κατανόησα από τη μετάφραση των όσων ε, διαβάσατε. Κατάλαβα καλά ότι λέτε ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε το πλαίσιο αποδοτικότητας να οριστεί καλύτερα, διότι Υπάρχει μεγάλος πειρασμός βέβαια για τις χώρες μέλη και εγώ ήμουν μέλος ε, Περιφερειακού Κοινοβουλίου όταν έρχονται λεφτά από τις Βρυξέλλες προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε τα δικά μας τα λεφτά, να τα βάλουμε κάπου στην άκρη. Αν κάποιος περνάει δίπλα μου με ένα σακί λεφτά προσπαθώ να πάρω κάτι κι εγώ. Άρα, το πλαίσιο απόδοσης. Για ποιο λόγο υπήρχαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και για ποιο λόγο όχι, αυτό δεν ήταν ξεκάθαρο ορισμένο. Αυτό λέτε εσείς. Ε, επ' αυτού λοιπόν πρέπει να εγκύψουμε. Να δούμε δηλαδή η τεχνική συνδρομή για ποια πράγμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε και για ποια όχι. Για τη δεύτερη έκθεση κάτι δεν κατανόησα και τόσο καλά. υπερκεφαλαιοποίηση, πλέον ή μάλλον υπερβολική κεφαλαιοποίηση των ταμείων χρηματοδότησης. Αυτό λέτε είναι καλό ή κακό οι Υπουργοί Οικονομικών θα σα πούν «Α, δόθηκαν πολλά λεφτά, εάν δεν απορροφηθούν θα τα πάρω πίσω». Αυτή είναι η πρόθεση, αυτό θέλω να μάθω. Ω πολιτικοί που ασχολούμαστε με τα γεωργικά πρέπει να φροντίζουμε βεβαίω να απορροφώνται σωστά τα κονδύλια. Δεν επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα μόχλευση, είπατε επίση. Μήπω οφείλεται, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Βρήκατε και καλά θετικά παραδείγματα, δηλαδή που σε ποια έργα επιτέθηκε πραγματικό αποτέλεσμα απόδοσης, αποτέλεσμα μόχλευσης. Βέβαια αυτά είναι κάπως νέα πράγματα και παλιά λέγαμε, κοιτάξτε, λεφτά υπάρχουν, κάνουμε, ε, προχωρούμε σε σχεδιασμό προγραμμάτων ε, επιδοτήσεων και αυτό είναι όλο. Τώρα προσπαθούμε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Να δούμε λοιπόν πώ γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι ακόμα καλά ορισμένο. Τέλο, μια παρατήρηση. Για μα τα χρηματοδοτικά εργαλεία στον χώρο της υπαίθρου είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Γνωρίζουμε ότι ο χώρος της υπαίθρου έχει διαρθρωτικά προβλήματα, αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα και γι' αυτό με στενοχωρεί όταν λέτε ότι διατέθηκαν χρήματα, μεν, ή εμείς διαθέσαμε χρήματα τέλος πάντων, αλλά δεν απορροφώνται. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Υπάρχουν και καλά παραδείγματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Διότι έχουμε αρκετές περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ακόμα μεγάλο δρόμο να καλύψουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου και για την παρουσία και για την παρουσίαση. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω κάποιες ε, πτυχές για τις οποίες ε, χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσει ε, και την άποψη για τα ζητήματα που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Ήμουν στην περιφερειακή κυβέρνηση και έχω και εγώ κάποια εμπειρία. Μιλήσατε για την τεχνική βοήθεια. Και είπατε ότι ίσως αυτές οι ενισχύσεις ε, ή δεν είναι επαρκείς ή δεν είναι καλά καθορισμένες και κατά την άποψή σας, αν κατάλαβα καλά, και θέλω να το ξεκαθαρίσετε, ε, είχαν ε, συνοδευτεί με πολλές δημόσιες δαπάνες Άρα, στο προηγούμενο, στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, 7-13 αναλύσατε, ουσιαστικά διατήρησαν κατά την άποψή σας ε, υπερβολικό βάρος ότι αυτό το διοικητικό, τα διοικητικά έξοδα διαχείρισης. Δεν είναι ότι απαγορεύεται αυτό βέβαια, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι δεν είναι ας πούμε η καλύτερη μορφή ε, δαπάνη των ε, χρημάτων αυτών που υποτίθεται προορίζονται καταρχήν για τεχνική βοήθεια, τεχνική συνδρομή. Άρα πρέπει να βρούμε μια ε, άλλη φόρμουλα. κατάλαβα καλά, στα περισσότερα κράτη-μέλη συνέβη αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι, μήπως δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, θεωρητικά, αυτή η τεχνική συνδρομή, ενισχύσει, δεν είναι ξεκάθαρα δηλαδή τα πράγματα και μήπω δεν είναι και ξεκάθαρε οι δαπάνε του πρώτου, ε, δεν υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ δαπανών πρώτου και δεύτερου πυλών. Και για το χρηματοπιστωτικό κανονισμό, κατάλαβα καλά, είπατε ότι αυτά τα μέσα δεν λειτουργήσαν καλά ούτε και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, γιατί αυτά τα εργαλεία, αυτά τα μέσα, τι είχαν ως βασικό στόχο, να προσελκύσουν νέα ιδιωτικά κονδύλια. Επειδή δεν υπήρχαν. Και έτσι να ε, δοθεί μεγαλύτερος προϋπολογισμός για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπέθρου Αυτό θα ήταν το ιδεώδης. Αναλύουμε όμως την περίοδο 7-13 με μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση που έπληξε τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα στη χώρα μου ήταν τεράστια η κρίση. Άρα δεν υπήρχαν δυνατότητες ουσιαστικά. για να προσελκυστούν νέα κεφάλαια ιδιωτικά για αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Πέραν της διαγύρισης θα δούμε αν ήταν επαρκής ή όχι. Θα μπορούμε να το κρίνουμε αυτό ίσως κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω ότι ο οικονομικός κύκλος, η χρηματοπιστωτική κρίση, η δημοσιονομική, η οικονομική κρίση που βίωσε η Ευρώπη και την ζήσαμε στη χώρα μου, στην Ισπανία και τη ζούμε, δεν βοήθησε στην δημιουργία ιδιωτικών κεφαλαίων που θα μπορούσαν να δώσουν όθηση και περισσότερο υπερπολογισμό στα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Και μια κριτική, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι ουσιαστικά χρηματοδότησαν τις επιδοτήσεις. Μα δεν υπήρχαν ε, δυνατότητες χρηματοδότησης επιδοτήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Εάν πάρουμε ένα στιγμιότυπο, αν θέλετε, φωτογραφικό, δεν είναι ε, κάτι που θα αντικατοπτρίσει την κατάσταση, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των αναγκών στο γεωργικό κλάδο. Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία συμπλήρωσαν ουσιαστικά τις επιδοτήσεις που είχαν δοθεί. αλλά δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλε περιπτώσει. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι πολλά οφείλονται στον οικονομικό κύκλο και σε αυτή την κρίση που βιώσαμε. Θα τα πείτε κι εσεί βέβαια καλύτερα. Θα μα δώσετε τη δική σα ερμηνεία και τη δική σα άποψη που θεωρώ πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι δύο αυτές ε, εκθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνουμε αυτή τη στιγμή, με από τις εκθέσεις αυτές, ότι ε, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικά και είναι ιδιαίτερα δαπανηρά. Οι περισσότεροι ενδεχομένω να το γνωρίζουν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσει λοιπόν τις πρακτικές της, τις παράλογες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μέσα τα οποία επηρεάζουν τελικά τις τελικές τιμές και βλέπουμε ότι αντί να χρησιμοποιήσουμε τελικά κάποια συγκεκριμένα μέσα, χρησιμοποιούμε όριστε πολιτικέ όσον αφορά την άπτυξη τη υπαίθρου. Βλέπουμε ότι τα τελικά αποτελέσματα δεν υπάρχουν καν τη στιγμή που οι γεωργοί μα, οι αγρότε μα βρίσκονται σε απόγνωση και βλέπουν ότι στην πράξη τίποτα συγκεκριμένο δεν γίνεται προκειμένου να εξαλειφθεί η κρίση την οποία γνωρίζουν αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά σκανδαλώδε και νομίζω ότι πραγματικά χρειάζεται μια έντονη αντίδραση από εμά, τα μέλη τη Επιτροπή Άγκρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Αφού αναλύσουμε τις εκθέσεις, πιστεύω ότι θα προκύψουν και άλλες απορίες που θα μπορούσαμε να σας θέσουμε είτε προφορικός είτε γραπτός και να λάβουμε αντιστοίχως και απαντήσεις. Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικά εργαλεία και χρηματοδότηση δημόσιο και ιδιωτικού τομέα και καλά αποτελέσματα βέβαια. Είπατε ότι δεν είχατε τη δυνατότητα να ελέγξετε κατά πόσο δόθηκε σωστά η τεχνική βοήθεια. Δεν ξέρω, μήπως δεν κατάλαβα πολύ καλά, αλλά αν δεν κατάλαβα καλά και δόθηκε τελικά σωστά η τεχνική βοήθεια. Θα πρέπει να δούμε μήπως ε, δεν εφαρμόστηκαν οι σωστές διαδικασίες ή δεν επελέγει η σωστή μεθοδολογία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πού εντοπίστηκαν τα προβλήματα. Έλλειψη χρόνου ήταν το θέμα. Έλλειψη πόρων. Και εγώ έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλος και είχα τη δυνατότητα να εφαρμόσω σε μια από τις περιοχές, σε μια από τις περιφέρειες, ένα πρόγραμμα ανάπτυξη πέθρου. Η Λιθουανία ήταν στο κύμα των ε, προσχωρήσεων το 2004 και για μας τότε ήταν ε, ε, η πρώτη τετραετία εκεί μέσα στο 7-13 χρειάστηκε να μάθουμε πολλά. Και να συνειδητοποιήσουμε το πώς πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα. Έπρεπε να κατανοήσουμε όλες τις λεπτομέρειες και να δούμε πώς θα μπορούσαμε με αυτή τη χρηματοδότηση να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Προσπαθήσαμε να προσελκύσουμε ιδιωτικούς επενδυτές. Και πρέπει να μπορώ να σας πω ότι στην Ήπεθρο Η αναλογία 50-50 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ζουν σε αγροτικές περιοχές και έχουν κονδύλια τα οποία μπορούν να επενδύσουν σε κάποια επιχείρηση. Δεν διαθέτουν πολύ απλά τέτοια κεφάλαια. Ζητήσαμε λοιπόν άδεια η αναλογία να είναι 65-35 Δηλαδή 65 από τα ταμεία και 35 από τον ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί και στο μέλλον αυτή η δυνατότητα, διότι υπάρχουν περιοχές όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και εκεί ε, θα μπορούσε να ισχύσει αυτή η διαφορετική αναλογία αντί του 50-50. Κάτι ακόμη, μπορώ να πω ότι χρειάστηκε να περιμένουμε για πολύ καιρό μέχρι να λάβουμε τα χρήματα. Και αφού είχε ολοκληρωθεί η σχετική εργασία ή το σχετικό έργο. Ίσως τα κράτη-μέλη καταχρώνται ενίοτε των καταστάσεων, δηλαδή παίρνουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλα ταμεία, αλλά αυτά τα χρήματα δεν τα δίνουν στους δικαιούχους, τα διατηρούν για μισό χρόνο, ένα χρόνο και πραγματικά υποφέρουν οι δικαιούχοι στο μεσοδιάστημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό το φαινόμενο και να φροντίσουμε άπαξ και το κράτος μέλος παίρνει τα χρήματα να τα δίνει αμέσως δικαιούχους. Ευχαριστώ. Έχω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω, δύο αιτήματα. Λαμβάνουμε κάθε μέρα πολλά έγγραφα αλλά σπάνια βλέπω τόσο καλά διαρθρωμένα και διατυπωμένα έγγραφα και με πάρα πολύ καθαρές δηλώσεις και εξυπηρετούν και ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν απαραίτητα τόσο καλά τα τεχνικά αυτά θέματα. Πρόκειται λοιπόν για πραγματικά θαυμάσεις εκθέσεις και πολύ χαίρομαι που δεν ε, τα λέτε αόριστα, διότι λέτε καθαρά ότι όταν πρόκειται για χρήματα που δαπανώνται, για παράδειγμα, για την συντήρηση δικτύων μηχανογράφησης ή για άλλα σχετικά, στην ουσία δαπανώνται για σκοπούς ξένους προς αυτούς για τους οποίους εγκρίθηκαν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις εκθέσεις αυτές, κυρίως για την πρώτη. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εκεί όπου λέτε συστάσεις, γράφετε μια φράση. Τι σημαίνει ακριβώς, λέτε μια φράση, ότι ενδεχομένως η πολιτική θα πρέπει να σκεφτεί η πολιτική με δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτεί και την ενδεχόμενη εγκατάλειψη των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων. Είναι στη σαλάδα 40 η σύστασή σας υπαριθμών 6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέτε θα πρέπει να προβληματιστεί, να λάβει υπόψη και το ενδεχόμενο της εγκατάληψής τους. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως μας συστήνει προτείνεται να διαγράψουμε απολύτω τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πάντω, επαναλαμβάνω τι ευχαριστίε μου και για τι δύο εκθέσει που υποβάλλατε. Σέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για τις δύο αυτές εκθέσεις και να πω ότι Ε, σωστά εστιάζουν στο κατά πόσον τα χρήματα δαπανήθηκαν λίγο πολύ σωστά με βάση τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως εγώ ε, θα ήθελα να δούμε ουσιαστικά και να συζητήσουμε αυτά τα χρήματα έχουν ε, θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο για τους αγρότες και για την υπεθρό. Μιλάμε για τεχνική βοήθεια. Τελικά μιλάμε για δημόσιο χρήμα, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει για την τεχνική βοήθεια, αλλά ε, με κακό τρόπο ουσιαστικά υποκαθίσταται η τεχνική βοήθεια που δινόταν από δημόσιους οργανισμούς, δημόσιους φορείς και δημόσιους κυβερνητικούς οργανισμούς. Άρα αυτό είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι πράγματι αποτελεσματικό με δημόσιο χρήμα να δημιουργούμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη γεωργία για τους αγρότες, τις αγρότησες, αλλά να διαλύουμε τις δημόσιες υπηρεσίες που παρήχαν οι κυβερνήσεις. Διότι τελικά αυτό που πάντα έχουμε είναι επισφαλείς ε, θέσεις ε, και συνθήκες εργασίας και χειρότερες δημοσίες υπηρεσίες. Για τη χρηματοδότηση τώρα το ίδιο. Ε, θα πρέπει να δούμε τα χρήματα δίνονται για τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας ή μήπως προωθείτε ε, ή μάλλον προωθείται τελικά αυτή η βιώσιμη αγροτική δραστηριότητα. Δεν νομίζω ότι γίνεται το ένα ούτε το άλλο. Η αποστολή του ελεγκτικού συνεδρίου είναι με τα πρότυπα και τους κανόνες που έχουμε να διαπιστώνει αν τα πράγματα γίνονται σωστά ή όχι, καλά ή κακά. Αλλά θα πρέπει εμείς ως Επιτροπή να δούμε και το πολιτικό σκέλος, να πάμε πιο βαθιά στο πολιτικό σκέλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ και εγώ να ευχαριστήσω για την υποβολή αυτή τη εκθέσεως που περιλαμβάνει πολλές κριτικές παρατηρήσεις. Έχω ωστόσο μια ερώτηση για τα ε, γραφήματα που έχετε στη σελίδα 16 και όπου αντιπαραβάλλεται την δαπάνηση των χρημάτων το 2007 με το 2013. Η διαδικτύωση έχει αναέβει τώρα στο, 18%, στο 28% συγγνώμη, Αναρωτιέμαι όμως αυτή η διαδικτύωση τι προσφέρει στον κόσμο που ζει στην Ήπεθρο. Είναι σωστή η χρήση αυτών των ε, κονδυλίων ε, στον τομέα αυτό. Επίσης αναφέρεστε επικριτικά στην διάθεση των προγραμμάτων, των ε, κονδυλίων μάλλον, σε διοικητικέ δαπάνε. Σωστό. Στη σελίδα 21, στην παράγραφο 47, λέτε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των χωρών μελών για την ε, συνολική χρηματοδότηση του ΕΛΑ για την τεχνική συνδρομή, τόσο λιγότερα κονδύλια κατευθύνονται τελικά σε έργα υποδομών στις, ε, στην Ήπεθρο. Δεν φαίνεται καθαρά ποια κονδύλια κατευθύνονται στη τεχνική συνδρομή και πόσα κατευθύνονται πραγματικά για τα μέτρα επενδύσεων στον χώρο της υπαίθρου. Σύμφωνα με την έκθεση, νομίζω ότι θα πρέπει εν πάση περιπτώσει στην Επιτροπή Γεωργίας να εγκύψουμε ξανά στο θέμα και να σκεφτούμε εάν αυτού του είδους η χρηματοδότηση μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πριν το πράξω αυτό, επιτρέψτε μου να θέσω κι εγώ ε, κάποιες ερωτήσεις και να τις συνοδεύσω με ορισμένα σχόλια. Ποιο ποσοστό του προϋπολογισμού για τα επιμέρους προγράμματα δαπανάτε κατά μέσον όρο για την τεχνική συνδρομή. Πώς κατανέμονται αυτά μεταξύ των νέων και των παλαιών χωρών μελών χρειάστηκε για τις νέες χώρες μέλη περισσότερη τεχνική συνδρομή σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας, για παράδειγμα. Υπάρχουν περισσότερα προγράμματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Υπάρχουν, είναι γνώμη μου, και είναι και πιο διαφοροποιημένα. Άρα υπήρχε και μεγαλύτερη ανάγκη ουσιαστικής στήριξης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η τεχνική συνδρομή είναι πολύ αναγκαία, παρόλο που υφίσταται συχνά κριτική διότι η τεχνική συνδρομή επιτρέπει την μεταφορά τεχνογνωσίας, know-how, που επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων. Ο ίδιος έχω εμπειρία σχετικά, διότι έχω ηγηθεί ενός σχετικού τμήματος στο παρελθόν και είναι σημαντικό να βρίσκεται κανείς σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει διότι πράγματι οι χώρες μέλη έχουν την τάση, αναφέστηκε ήδη αυτό, να βάζουν στη χρηματοδότηση αυτή διάφορους τομείς του προϋπολογισμού. Καμιά φορά υπάρχει βέβαια σχετική αναγκαιότητα, αλλά υπάρχει πάντα και δυνατότητα να συμφωνήσει κανείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον προβάλλει τα απαραίτητα, τα σωστά επιχειρήματα και εφόσον το αιτιολογήσει επαρκώς, το θεμελιώσει επαρκώς το αίτημα αυτό. σωστό θα είναι να προσληφθούν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες εδώ για να μπορέσουμε να να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από διάφορους, από την ε, τεχνογνωσία άλλων. Τώρα, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα ισχύσουν περισσότερα, περισσότερο από το ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο, δηλαδή επί μακρύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί το 1 συν 2 δεν αρκεί. Ως τώρα, για παράδειγμα σε έργα που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα, η Κομισιόν εποπτεύει της πρώτης ανακύκλωσης των κονδυλίων ενώ οι επόμενες φάσεις γίνονται σύμφωνα με την παλιά διαδικασία. Υπάρχουν, έχουν συλλεχθεί εδώ εμπειρίες και με διάφορες χρηματοδοτήσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι καλό που εξετάζουμε τώρα τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία και τα υλοποιούμε ως πιλωτικά προγράμματα. Τις δίνουμε λοιπόν τη μορφή με την οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο και στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Να δώσω τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να λάβουμε και εμείς μέρος σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχαριστήσω όμω και την κυρία Κάλιου Λάιντ για την παρουσίαση που έκανε και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για τι δύο πολύ ενδιαφέρουσε αυτέ ειδικέ εκθέσει, τι οποίε συνέταξε η, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και παρακολουθήσαμε εμεί με μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικά, όσον αφορά την πρώτη ειδική έκθεση, αυτή που έχει να κάνει με την τεχνική συνδρομή. Θα πρέπει να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και δέχεται μάλιστα και όλες τις συστάσεις του με μία μόνη εξαίρεση, στην οποία θα ήθελα να επανέλθω λίγο αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Προτού όμως περάσουμε τώρα στις συστάσεις που μας κάνατε, θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση, αν μου το επιτρέπετε, και το θίξατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, καθώς επίσης και άλλα μέλη της Επιτροπής σας τι είναι η τεχνική συνδρομή, τι είναι η τεχνική βοήθεια. Στα πλαίσια τη πολιτική, τη γεωργική και τη ανάπτυξη πέθρου, η τεχνική συνδρομή χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων και μπορεί να χρηματοδοτήσει και δραστηριότητε που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων των γεωργικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για μια στρατηγική προσέγγιση προκειμένου να ευοδοθούν τα προγράμματα και σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες τα κράτη-μέλη έχουν μια κάποια ευελιξία για το πώς χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική συνδρομή και είναι απαραίτητη η ευελιξία αυτή προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές διαφορετικές ανάγκες τις οποίες αντιμετωπίζουν στην πράξη κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών κατά την επιχειρησιακή φάση δηλαδή των προγραμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές τοπικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, στην περίοδο 2007-2013 είχαμε νέα κράτη-μέλη τα οποία για πρώτη φορά χρειάστηκε να εφαρμόσουν τη γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκε λοιπόν να υπάρχει μια κάποια ευελιξία προκειμένου να προσαρμοστούν με τις νέες απαιτήσεις τα νέα αυτά κράτη-μέλη και να εφαρμόσουν καλύτερα τα προγράμματα. Να περάσω τώρα στι συστάσει. Το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνική συνδρομή από τα κράτη-μέλη και να κάνει μία διάκριση ανάμεσα στο capacity building, δηλαδή της, τη χρηματοδότηση τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων και να γίνει μια διάκριση με τι διοικητικέ καθαρά δαπάνε. Εμεί δίνουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ προκειμένου όντω να γίνει αυτή η διάκριση και να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει στα κράτη-μέλη υποχρέωση αναφοράς των διοικητικών δεπανών ξεχωριστά, προκειμένου να φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η τεχνική συνδρομή και εντελώ ξεχωριστά ποιε είναι οι καθαρέ διοικητικέ δαπάνε. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε τελικά ποιε είναι οι επιδόσει αυτή τη τεχνική συνδρομή. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη στο μέλλον να μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες προκειμένου να βελτιωθεί η παρακολούθηση των δαπανών εκείνων που γίνονται στα πλαίσια της τεχνικής συνδρομής. Θα καταβάλουμε λοιπόν περισσότερες προσπάθειες με τα κράτη-μέλη για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σύσταση. Επίση, μα ζητά το ελεγκτικό συνέδριο να δημιουργήσουμε ένα ειδικό σύστημα παρακολούθησης για τεχνική συνδρομή και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση των αναγκών, καθώς επίσης και ένα μηχανισμό θέσης στόχων και παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών των στόχων. Σε μια πρώτη φάση εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τους απαραίτητους δείκτες για την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης τεχνικής συνδρομής. πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης τεχνικής συνδρομής προκειμένου να φαίνονται πραγματικά ποια είναι η συμβολή της τεχνικής συνδρομής στα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης. Και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται και σε μια ανησυχία που εξέφρασαν πολλά μέλη της Επιτροπής Άγκρη. Δηλαδή να γνωρίζουμε επακριβώς Πού πάνε τα χρήματα αυτά από τεχνική συνδρομή. Επίση, το λεκτικό συνέδριο μα ζητά να εγγυηθούμε ότι οι γενικέ διοικητικέ δαπάνε και ιδιαίτερα ότι οι δαπάνε συντήρηση των συστημάτων πληροφορική, συστήματα που χρησιμοποιεί τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη-μέλη, ότι οι δαπάνε αυτέ συντήρηση θα πρέπει να θεωρούνται συνήθει τακτικέ δαπάνε και να μπουν σε άλλη γραμμή του προπολογισμού. Τώρα εμείς εκεί έχουμε μία μικρή ένσταση και ποιο είναι το πρόβλημά μας κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι δαπάνες τεχνικής συντήρησης των συστημάτων πληροφορικής είναι δαπάνες συντήρησης εξελικτικές θα τις χαρακτήριζα. Δηλαδή προσπαθούμε να επικαιροποιούμε, να ενημερώνουμε τα συστήματα πληροφορικής. Με άλλα λόγια, πού είναι το πρόβλημα. Όταν εγώ το πρωί ανοίγω τον υπολογιστή μου και βλέπω στην οθόνη ότι υπάρχει μια προειδοποίηση η οποία μου λέει ότι κοιτάξτε η εκδοχή του λογισμικού που χρησιμοποιείται η 2,0 για παράδειγμα έχει επικαιροποιηθεί και έχει γίνει τώρα 3,0 αυτό για μένα δεν αποτελεί τακτική καθημερινή συντήρηση αλλά είναι ένα, μια εξελικτική αν θέλετε συντήρηση είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συνεχή χρονική βάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μας επιτρέπετε να περιλαμβάνουμε και τις δαπάνες αυτές στα πλαίσια της τεχνικής συνδρομής. Οι επικαιροποιήσει αυτές, η αναβάθμιση του συστήματος είναι πολύ σημαντική για την ίδια την υλοποίηση της τεχνικής συνδρομής. Αν οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να εγγραφούν στο γενικότερο προπολογισμό της τεχνικής συνδρομής, τότε πολύ φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα απαρχαιωθούν τα συστήματα αυτά της πληροφορικής και δεν θα είναι τελικά χρήσιμα. Όσον αφορά πάλι την τεχνική συνδρομή, να πω το εξή. Στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έχουμε προβλέψει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ένα μέγιστο 4% όσον αφορά τις δαπάνες για τεχνική συνδρομή. Αυτό είναι το νότατο όριο που έχουμε θέσει. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή προσπαθεί να παρακολουθεί με τρόπο συντηρητικό θα έλεγα τις δαπάνες που γίνονται στον τομέα αυτό και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεπεράσει το 1,16% ενώ έχουμε θέσει ως ανώτατο όριο το 4%. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι υπήρξε αύξηση της τεχνικής συνδρομής αλλά αυτό έγινε προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάποια νέα δίκτυα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υλοποίηση των προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης και για την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής που πρέπει να ανταποκριθούν αποκριθούν σε μια νέα νομοθεσία που χρησιμοποιεί κατά ευρύτερο τρόπο και πολύ περισσότερο τα συστήματα πληροφορικής. Νομίζω λοιπόν ότι η χρησιμοποίηση των κονδυλίων τεχνικής συνδρομής για αυτούς τους λόγους ήταν πολύ σωστή. Όσον αφορά τώρα τα χρηματοδοτικά μέσα και τη δεύτερη εκθεσή σας, ξέρετε ότι ε, είχαμε μία πρώτη πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το ζήτημα αυτό και ο Επίτροπός μας έχει δεσμευτεί πάρα πολύ για την ε, χρηστή χρησιμοποίηση και την ευρεία χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών αυτών μέσων όσον αφορά τα συστήματα πληροφορικής. Έτσι λοιπόν, βλέποντας την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, συντοποιούμε ότι μας δίνεται μια πολύ σημαντική ευκαιρία να δώσουμε μία νέα όθηση στις πρωτοβουλίες αυτές του Αρμοδίου Επιτρόπου. Τα χρηματοδοτικά λοιπόν μέσα μπορούν να αποτελέσουν, όπως σας είπα, μια πολύ σημαντική ευκαιρία, αλλά παράλληλα τα μέσα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο, παράλληλα με τα άλλα συστήματα, τα παραδοσιακά συστήματα επέμβασης για την υλοποίηση της γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσω των χρηματοδοτικών μέσων μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα, αρκεί όμω να υπάρχει και η πραγματική συνεργασία των κρατών μελών αλλά και των δικαιούχων. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη λοιπόν αυτή έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, δεχόμαστε όλες τις συστάσεις του συνεδρίου. και νομίζω απλώς ότι θα πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο τον προτινόμενο προπολογισμό για την περίοδο 2007-2013. Όπως είπε και η κυρία Αγγιλέρα, η περίοδος αυτή 2007-2013 είναι μια ειδική, ιδιαίτερη περίοδος. Δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποια θετικά αποτελέσματα γιατί διανύαμε μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση και επομένως πάρα πολλά έργα, πάρα πολλά προγράμματα δεν υλοποιήθηκαν, γιατί δεν το, δεν το επέτρεπε το γενικότερο αντίξω οικονομικό πλαίσιο. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα για πρώτη φορά. Και συνεπώς χρειάστηκε να περάσει μια περίοδος προσαρμογής για αυτά τα κράτη-μέλη προκειμένου να εξοικειωθούν καλύτερα με αυτά τα μέσα. Εμείς καταβάλουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να επιλύσουμε επιμέρους προβλήματα που έχουν προκύψει. Η πρώτη μας, αν θέλετε, προσπάθεια έχει να κάνει με τον ε, επανορισμό του νομοθετικού πλησίου και την εισαγωγή κάποιων νέων κανόνων. Ένας κανόνας, για παράδειγμα, είναι η εκ των προτέρων αποτίμηση των μέσων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη νέα περίοδο προγραμματισμού, 2014-2020 δηλαδή, Γίνεται λοιπόν μια υποχρεωτική εξάντεκ των προτέρων αξιολόγηση, προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς ποια χρηματοδοτικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν για ποια προγράμματα ακριβώς. Έχουμε συντάξει και ένα εγχειρίδιο για την καλύτερη χρησιμοποίηση αυτών των μέσων και στα πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου υπάρχουν πλέον κάποιες νέες διατάξεις που μας επιτρέπουν να αποφύγουμε όλα τα προβλήματα υπερκεφαλαιοποίησης τις οποίες στήξατε και εσείς και τις τα οποία είδαμε στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη χρησιμοποίηση αυτών των μέσων. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει πλέον στα κράτη-μέλη κάποιους νέους προσανατολισμού, μία δέσμη νέων προσανατολισμών, καθώς επίσης και κάποια βοηθητικά έγγραφα, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη καλύτερα και πιο αποτελεσματικά αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Τα έγγραφα αυτά απευθύνονται κυρίως στις δημόσιες διοικητικές αρχές. Όπως υπόθηκε και πριν από λίγο, υπάρχει όμως όντως ένα μνημόνιο κατανόησης με την, Παγκόσμια Τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Δημιουργήσαμε επίσης και μία πλατφόρμα, την BF Compass, η οποία θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως άλλωστε το είπε και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει τη χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Ο στόχος λοιπόν αυτός θα επιτευχθεί μόνο αν τα κράτη-μέλη και οι τελικοί δικαιούχοι το επιθυμούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όντως νομίζω ότι ήταν ε, πολύ θετικά αυτά τα οποία μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ε, παρέμβασή σας. Να ζητήσω τώρα από την εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να ξαναπάρει το λόγο και να απαντήσει σύντομα στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των ε, βουλευτών και του εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Στι ερωτήσει θα προσπαθήσω να απαντήσω στι περισσότερε, αν όχι όλε. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση ε, τη απόδοση τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, κυρίω Γιάρε την ερώτηση. Δεν έχει περιληφθεί στο πλαίσιο, στην αξιολόγηση των. Ε, το θέμα αυτό. Και είπα και στην παρουσίασή μου, το μισθολογικό κόστος αυτό που ε, διένυμαν ε, τα ε, γεωργικά κονδύλια και για τον πυλώνα 2 και για τον πυλώνα 1 δεν καλύπτονταν. Αν αυτό θεωρείται τώρα διοικητικές δαπάνες, αμυγός διοικητικές δαπάνες, ούτε λόγος, ούτε ανάγκη, ούτε δυνατότητα υπάρχει ανάλυση της επίδοσης. Πρέπει να είναι ξεχωριστό αυτό κατά την απόψή μου. Τώρα, καταρχήν δεν είναι δική μου δουλειά να πω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν μπορούν να πούν ότι πρέπει να καταβληθεί μόνο το μισθολογικό κόστος. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. 4% ας πούμε του προπολογισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου μπορεί να συμβάλλει και στην τεχνική βοήθεια και στο καθημερινό κόστος λειτουργίας ε, των ε, προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο αυτό η τεχνική βοήθεια προς το παρόν υποτίθεται ότι βοηθά τον κλάδο, πάντα και μόνο. Αυτό όμως δεν είναι διαφανές και αυτό ήταν ε, ο λόγος που με κριτική. Αν έχουμε πιο ξεκάθαρο ορισμό, και κάποιος είπε είναι μόνο για την εφαρμογή, όχι. Είναι νόμιμη η δαπάνη των ποσών αυτών για τεχνική βοήθεια. Απλά δεν θα πρέπει αυτή την τεχνική βοήθεια να την ε, θεωρήσουμε διοικητικό κόστος για την ανακεφαλαιοποίηση αν αυτό είναι καλό ή κακό. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ κακό, διότι αν όπως είπα, αν δούμε ότι 250 εκατομμύρια εγγυήσεις ε, είναι ένα ποσό το οποίο δόθηκε στους τελικούς δικαιούχους, ας υποθέσουμε ότι ένα στα πέντε έργα θα αποτύχει. Άρα έχουμε 20% ποσοστό κινδύνου, άρα πρέπει όλες οι εγγυήσεις ε, τελικά να καταβάλλονται ε, και πρέπει να έχουμε μία πρόβληση 50 εκατομμύρια 420 ήταν. Άρα 250 εκατομμύρια θα ήταν αν είχαν αποτύχει όλα τα σχέδια. Εμείς βάλαμε διπλό ποσό. Ε, σαν είχαν αποτύχει όλα τα προγράμματα δύο φορές δηλαδή. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα χρήματα δεν έχουν χαθεί. Κάθονται ε, στα ταμεία και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για καλύτερους σκοπούς. Επίσης αν υπάρχει ε, σοβαρή κρατική ανακεφαλοποίηση, γιατί κάποιος θα πρέπει να αναζητήσει ιδιωτική μόχλευση για ένα ε, τέτοιο ταμείο. Δεν γίνεται αυτό. Άλλη ερώτηση. Αν είχαμε στο κάποιο βαθμό μόχλευσης κάπου, ναι, στη Γαλλία στην ε, Κορσική και, στην Πούλια της Ιταλίας και στη Ρουμανία ε, προβλέφθηκε. Η Ιταλία και η Ελλάδα ήταν τα μόνα κράτη-μέλη όπου ρητός είχαν σχεδιαστεί τα ε, μέσα για μόχλευση στην Ελλάδα. Θα υπήρχε και η συμμετοχή των τραπεζών ως χρηματοδοτικός εταίρος, αλλά το Μάιο του 2014 δεν είχε επιτευχθεί κανένα αποτέλεσμα μόχλευσης. Άρα ακόμα και αν προβλεπόταν δεν επιτεύχθη. Technical assistance provided, uh, whether the court Τεχνική βοήθεια, αν μπορεί το ελληνικό συνέδριο να κάνει τη διάκριση μεταξύ της πραγματικής τεχνικής ε, βοήθειας αφενός και του κόστους ε, διαχείρισης αφετέρου. Ίσως, ναι, πράγματι, μπορούσαμε να δούμε στον έλεγχο πώς έγινε η διανομή της τεχνικής βοήθειας, αλλά δεν υπήρχε ροή αναφορών, άρα συνολικά δεν μπορεί να πει κανεί ότι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναλογία τάδε τη τεχνική βοήθεια πήγε σε καθημερινό κόστο διαχείριση και ότι αυτό προωθεί την τομεακή ανάπτυξη. Οι δυσκολίε ε, για να φανεί τελικά τι δαπανήθηκε και πού, κυρίω στο το θέμα ε, της επιλεξιμότητα, γιατί τα κράτη-μέλη έπρεπε να αποφασίσουν και να αποδείξουν ε, ότι τα χρήματα πήγαν για τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2. Τεχνική βοήθεια όμως αυτή προβλεπόταν για τον πυλώνα 2 μόνο. Βέβαια υπάρχουν καταστάσεις όπου τα ίδια άτομα εργάζονταν και για τους δύο πυλώνες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να γίνει ανάλυση. Αυτά ε, διαπιστώσαμε. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών, αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα κάνουμε μια γενική ανάλυση ως ελεγκτικό συνεδρίο των καθυστερήσεων πληρωμών σε τις εκθέσεις μας, άρα μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία εκεί. Είναι όμως μια γενική ανάλυση. Τι δεν έχει καταβληθεί από την Κομισιόν σε επίπεδο κρατών μελών, αυτό γίνεται από τα κράτη-μέλη, όχι για το, ε, δεν το, το αναλύουμε εμεί ω ελεγκτικό συνέδριο αυτό το θέμα. Τώρα, για τη σύσταση 6, ε, στρατηγική εξόδου δηλαδή, από το Ταμείο και τα χρηματοπτικά μέσα του Ταμείου Ανάπτυξη Πέθρου. Θεωρούμε ότι το Ταμείο δίνει εγγύησει. Και λύγει κάποια στιγμή, στο τέλο του περίοδου προγραμματισμού. Και εκεί πρέπει να υπάρξει διαδικασία κλεισίματο. Οπότε το Ταμείο κλείνει. Και τα εναπομένοντα χρήματα διανέμονται σε άλλα μέτρα. Ή μπορεί να συνεχιστεί να ισχύει και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού οι κανόνες περί κλεισίματος δεν μου είναι και ιδιαίτερα ξεκάθαροι και θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δω ποιος είναι ο συντελεστής στον οποίο ε, γίνεται αποδεκτό ως, γίνεται αποδεκτή ως δαπάνε αυτό ε, το κόστος. Στο, στην περίπτωση της ανακεφαλαιοποίησης υπάρχει κάποιο περιθώριο για να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα. Αν οι δηλαδή θεωρούνται κόστος ή όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις η Κομισιόν θεωρεί κόστος. Επίσης τα χρηματοδοτικά μέσα κάποια κράτη-μέλη δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορούν να τα μεταφέρουν στην άλλη περίοδο. Είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα αυτό τώρα. Σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια, έχουμε τα δίκτυα, τα γεωργικά δίκτυα, Rural Networks. Ένα άλλο θέμα ήταν ένα γράφημα για την τεχνική βοήθεια ε, για τις δαπάνες ε, τεχνικής βοήθειας σε επίπεδο κομισιών και μία μικρή διαφωνία, η μόνη που έχουμε σε τεχνικό επίπεδο με την κομισιόν. Εμείς ε, ομαδοποιημένα βλέπουμε ότι επιχειρησικές και μη επιχειρησικές δαπάνες από το 7 έως 13, από το 12 πήγανε σε 22 εκατομμύρια και βλέπουμε επίσης ότι μειώθηκε ο προπολογισμό από 12 σε 8 και είδαμε ότι οι διαθέσεω πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν επιτρέπουν να κατά. Development. Uh, και το μη επιχειρησιακό κόστος πληροφορικής φαίνεται να χρηματοδοτείται περισσότερο. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την κριτική. Ενώ οι διοικητικοί προπολογισμοί συρρυκνούνται σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο κομισιών, αυτό που ε, μετράς, αυτό βλέπεις τελικά. Απλά κάποιε φορές μπορεί να βλέπεις και αύξηση κάπου αλλού. Αλλά ουσιαστικά περί του ίδιου πρόκειται. Τώρα, ποσοστό τεχνικής βοήθειας, ε, ο μέσος όρος για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού ήταν λίγο κάτω από το 2% ε, και από το 0,99% το 4% ε, διακυμάνθηκε στο πλαίσιο του προπολογισμού ανάπτυξης της υπαίθρου. Κάποια κράτη χρησιμοποίησαν περισσότερο, κάποια λιγότερο αυτό το προπολογισμό. Υπάρχει μια τάση να αυξηθούν τα ποσά. Και υπάρχει ένα παράρτημα, αν θέλετε να δείτε, σε κάθε κράτος μέλος, σελίδα 37 της έκθεσης, το παράρτημα αυτό, ένα πίνακα δηλαδή, με κατανομή και με νούμερα συγκεκριμένα για κάθε κράτος μέλος. Τα χρηματοδοτικά μέσα, τι πρέπει να υπηρετούν, πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται. Κάποιος είπε ότι εμείς προτείνουμε να κλείσουν αφού είμαστε τόσο αρνητικοί. Όχι, δεν προτείνουμε κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Θεωρούμε στο Ελληνικό Συνέδριο ότι τα χρηματοδοτικά μέσα ουσιαστικά σημαίνουν ότι μπορούν τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν πάνω από μια φορά. Να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα δηλαδή. Αυτή η αρχή πρέπει να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά. Άρα ο στόχος να έχουμε περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα, διπλασιασμό σε σχέση με την προηγούμενη δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα στόχος ώστε η μόχλευση και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επιτυγχάνονται και δεν είμαστε βέβαιοι ότι το νέο πλαίσιο προγραμματισμού αυτομάτως πετυχαίνει αυτούς τους σκοπούς. Χρειάζεται λοιπόν να παρακολούθησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάντα σημαντικό ε, να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων, από την οποία φάνηκε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την επικοδομητική αυτή συνεργασία που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Η εργασία που κάνει το Ελεκτικό Συνέδριο είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τις δικές μας εργασίες. Και παράλληλα μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε με τη δική μας τη δουλειά, τονίζοντας κάθε φορά τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής πολιτικής. Μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή και εμείς από τη δική μας την πλευρά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο προκειμένου να ερμηνεύει καλύτερα τις δαπάνες που γίνονται στα πλαίσια του γεωργικού τομέα. Εκτιμούμε πάντως πάρα πολύ την εργασία που κάνετε στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Όπως σας είπα, ευελπιστούμε να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή που έχουμε και θα θέλαμε να έχουμε και άλλες παρουσιάσεις στο μέλλον. Ο κύριος Γιάρπαλη θέλει το λόγο. Πολύ σύντομα, επειδή θα γίνει μετά συνάντηση των συντονιστών, έχω έτσι αυθόρμητα μια ιδέα. Να ορίσουμε έναν διαρκή εισηγητή. Θεωρώ τον διάλογο με το ελεγκτικό συνέδριο πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να μπορεί ωστόσο η συζήτηση αυτή να μπαίνει και σε λεπτομέρειες που δεν είχαμε την ευκαιρία, δεν είχαμε τον χρόνο δηλαδή σήμερα. Μαζί με τους συντονιστές να βρούμε λοιπόν ένα τρόπο να διεξάγουμε διαρκή διάλογο. Δηλαδή να συναντιόμαστε συχνότερα με την εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου και να συζητούμε περισσότερο και συχνότερα και σε βάθος. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος. Όντως, καλή ιδέα. Είναι πολύ καλή ιδέα. Θα επιτρέψει έτσι και έναν διαρκή και περισσότερο σε βάθος προβληματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Καριουλάιτ. Εκφράζω ξανά την ελπίδα να συνεχιστεί η συνεργασία που είμαι βέβαιος ότι θα είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές, δηλαδή και ε, για σας και για μας, αλλά και κυρίως για την Γεωργία και την Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Είστε πολύ ενθαρρυντικοί. Θα τα μεταφέρω στους συναδέλφους μου. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ας περάσουμε λοιπόν ευθύ αμέσω στο σημείο 6 της μερίσιας διάταξης. Θα το παρουσιάσω εγώ αυτό το σημείο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε τον καθορισμό ανωτά του ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέους στα έλια και τα λίπη και θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδια... αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης. Λοιπόν, αναφερόμαστε εδώ πέρα στον κανονισμό 320 κάθετος 2006 και ακολουθούμε το άρθρο 50 του κανονισμού. Ουσιαστικά μας ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσουμε δύο κείμενα τα οποία είναι πλέον παροχημένα. Και κατά αυτόν τον τρόπο τόσο ο κανονισμός όσο και οδηγία θα είναι πιο αποτελεσματικά και πιο διαφανή. Έχουμε λοιπόν την οδηγία 76 621 όσον αφορά τον καθορισμό ανώτατου ορίου περιεκτικότητας ερωτικού οξέως, τα έλε και τα λύπη, καθώς επίσης και τον κανονισμό 320-2006 για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος στην αδιάρθρωση του κλάδου της ζάχαρης. Στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου οι συντονιστές ζήτησαν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκριθεί χωρίς τροπολογίες και με την απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού μας. Αποφάσισα λοιπόν εγώ να προετοιμάσω και να παρουσιάσω την έκθεση αυτή στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας σας έδωσα κάποιες προκαταρκτικές πληροφορίες. Η έκθεση που παρουσιάζω σήμερα ουσιαστικά σας ζητά να αντικατασταθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εγκριθεί από τη νέα της πρόταση χωρίς να υποβληθούν τροπολογίες. Οι δύο πράξεις που αναφέρθηκα έχουν καταστεί πλέον παροχημένες, επομένως στην πράξη δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο. ουσιαστικά έχουν ενσωματωθεί, έχουν απορροφηθεί η οδηγία και ο κανονισμό σε άλλες νομοθετικές πράξεις. Γι' αυτό το λέω ότι έχουν καταστεί παροχημένες οι νομοθετικές αυτές πράξεις. Και ζητήθηκε μάλιστα από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου να γίνει μια αλλαγή στη νομική βάση με αναφορά πλέον στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την χρήση του ερκικού οξέως. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού μας για αλλαγή νομικής βάσης, πρέπει η Επιτροπή Γιούρι, νομικών θεμάτων δηλαδή, να υποβάλει μια γνωμοδότηση, προκειμένου να μας πει αν όντως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα αυτή νομική βάση την οποία προτείνει το Συμβούλιο. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με την καθήλυνα αυτήν αρμόδια Επιτροπή, την Επιτροπή Γιούρι, και τη ζητήσαμε να συντάξει και να υποβάλει γνωμοδότηση. Δεν προβλέπονται λοιπόν εξημών τροπολογίες, μολονότι υπάρχει επίσημη ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών, θεωρητική βέβαια. Είναι 23η Ιουλίου του 2015. Έχουμε τον αναπληρωτή διευθυντή της DG Agri μαζί μας. Να ζητήσω λοιπόν από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο, προκειμένου να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το ζήτημα αυτό. Ας είμαστε όμως σύντομοι, παρακαλώ πολύ. Ενδεχομένως, ε, κύριε Διευθυντά, αν υπάρχουν ερωτήσεις, να μπορέσετε να απαντήσετε και στη συνέχεια, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα. Thank you, Chairman. I can be very, very brief. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Υποστηρίζουμε απολύτως το σχέδιο εκθέσεως που έχετε καταθέσει. Έχει τεχνικό χαρακτήρα με την έννοια ότι δύο νομοθετήματα τα οποία έχουν πλέον απολέσει την ουσιαστική τους ισχύ θα πρέπει να διαγραφούν ώστε οι πολίτες όταν αναζητούν όταν εξετάζουν το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουν απέναντί τους απερχαιωμένα νομοθετήματα. Όντω το άρθρο 114 της ε, συνθήκης είναι η σωστή βάση ε, θεσπίζει κοινή αγορά. Έχει λοιπόν οριμάσει ο χρόνος για να προχωρήσουμε με αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο πρόεδρος Έχετε καμιά ερώτηση εσεί οι βουλευτέ. Όχι. Καλά λοιπόν. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται η πρόταση. Εάν υπάρξουν τροπολογίε δεν σας καλώ να υποβάλλετε τροπολογίε, αλλά εάν υπάρξουν, όπως είπα, η προθεσμία λήγει στι 23 Εβδόμου. Αναμένουμε και τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, μετά θα συζητήσουμε ξανά και μετά θα καταλήξουμε στην Ολομέλεια. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά και ε, προχωρώ στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ανταλλαγή δηλαδή απόψεων με προσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρα για την καταπολέμηση της διασυνοριακής Εξάπλωση της αφρικανικής πανόλης των χείρων, καθώς και για τι επιπτώσει της στον γεωργικό τομέα. Οι επιπτώσει του γεωργικό τομέα βεβαίω είναι σημαντικέ, αλλά και η μετακίνηση των ορίων εξάπλωσης της νόσου, ε, που αποτελεί κίνδυνο. Χρειάζεται αύξηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών καταπολέμησης και να είμαστε σε θέση να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ενδεχόμενο κίνδυνο εφόσον αυτό εμφανιστεί. Και εκεί απαιτείται μια ε, σοβαρή προετοιμασία. Έχουμε προσκαλέσει εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας πληροφορήσουν. Πρόκειται για νόσο η οποία προκαλεί μεγάλες καταστροφές. Πρόκειται για μολυσματική νόσο, δεν υπάρχουν και εμβόλια που να επιτρέπουν την αντιμετώπιση του ιού, οι βαλτικές χώρες και η Πολωνία σημείωσαν κάποια κρούσματα της νόσου το 2014, εν ώψη δε του γεγονότος ότι υπάρχει υπόνοια ότι η νόσος φτάνει μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία και από τη Λευκορωσία, τίθεται το ερώτημα τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει, ώστε να μπορέσει να αναλύσει την εξάπλωση της νόσου και πώς σχεδιάζει να συνδράμει τους κτηνοτρόφους. Διότι η νόσος έχει βεβαίως και βαρύτατες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή και στην προμήθεια κρέατος στην αγορά. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τον κύριο Βαν Ρούτεμ να λάβει το λόγο. Έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε εσείς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω λίγο την παρουσίασή μου αυτή χρησιμοποιώντας το PowerPoint το οποίο βλέπετε και στις οθόνες σας. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι ε, το ζήτημα αυτό της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων αφορά πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο την προηγούμενη εβδομάδα στο Βίλνιους συναντήθηκαν οι Υπουργοί Γεωργίας προκειμένου να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και να δούνε πώς μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νόσου αυτής. Να σας πω καταρχάς ότι η Αφρικανική Πανόλη των Όλων εξαλείφθηκε από κάποια άλλα κράτη-μέλη. Βλέπετε εδώ πέρα στην οθόνη σας διάφορες ημερομηνίε κατά τις οποίες κράτη-μέλη κατάφεραν να εξαλείψουν, να εξαφανίσουν αυτή την ασθένεια. Δεν καταφέραμε όμως να εξαλείψουμε την ασθένεια στην Σαρδινία εξαιτίας της τοπικής ε, κατάστασης είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις των αγριόχειρων. Λοιπόν, μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Οι επιδημολογικές έρευνες καταδεικνύουν ότι το 2007 πέρασε στη Γεωργία η νόσος αυτή, μέσω πλοίου από τη Μοζαμβίκη και πραγματικά περνάω τώρα πάρα πολύ γρήγορα τις διαφάνειες μόνο και μόνο για να σας δείξω πώς έφτασε τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος αυτή, η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Βλέπετε στη συνέχεια του 2007-2009 στη Γεωργία πώς εξελίχθηκε η νόσος αυτής. Αυτή περνάμε στο 2011 και φτάνουμε τελικά στο 2014 όπου βλέπετε εδώ πέρα τις αιστείες της νόσου αυτής στη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία. Και το 2014 είχαμε και το πρώτο κρούσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε καθαρά στατιστική βάση, στη διαφάνεια αυτή, βλέπετε την καταγεγραμμένη εμφάνιση της νόσου στους άγριους χείρους στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας, στην Ρωσία, στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπετε κάποια κρούσματα τα οποία βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως βλέπετε ξεκάθαρα στο χάρτη αυτό, στην Λευκορωσία δεν είχαν κοινοποιηθεί κάποια κρούσματα προς τον παγκόσμιο οργανισμό, το, μάλλον το γραφείο επιζωτιών, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι δεν υπήρξε διαφάνεια από πλευράς των αρχών της Λευκορωσίας. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα γύρω από τη Λευκορωσία, αλλά όχι στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε εδώ με τις κίτρινες κουκίδες τις περιπτώσεις εκείνες εμφάνισης της νόσου στα αγριογούρουνα, τα οποία βρέθηκαν νεκρά και στα οποία διαγνώστηκε φρεκανική πανόλη των χείρων, αλλά καταφέραμε να απομονώσουμε την νόσο με τους αστερίσκους βλέπετε κρούσματα σε συγκεκριμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Με την εξαίρεση δύο μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όλα τα, όλα τα υπόλοιπα κρούσματα εμφανίστηκαν κυρίως σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, όπου χείροι είχαν έρθει σε επαφή με αγριογούρουνα. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε κάποια κρούσματα στα σύνορα με την Εστονία και την Λετονία, και βλέπετε ότι τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία. Τώρα, ποια είναι τα μέτρα αυτά τα οποία αποφάσισαν να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε μια πλήρη εναρμόνιση της ατμοτροφικής νομοθεσίας, η οποία δεν είχε επικαιροποιηθεί από τη δεκαετία του 80. Έχουμε επίσης συγκεκριμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης, εθνικά σχέδια αυτά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση αφρικανικής πανόλης των χείρων. Είχαμε επίσης ε, τη χρησιμοποίηση ενός σημαντικού ευρωπαϊκού εργαστηρίου αναφοράς όσον αφορά την αφρικανική πανόλη των χείρων και μας βοήθησαν στα πλαίσια της διάγνωσης και διάφορα εθνικά εργαστήρια αναφοράς. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτήσαμε τα μέτρα έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης και τα προγράμματα εξάλληψης και πέρα από την αντιμετώπιση τη αυτής αυτή καθ' προχωρήσαμε επίσης και σε κάποια προγράμματα, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, προκειμένου οι πολίτε να γνωρίζουν πώς έχει κατάσταση. Χρησιμοποιούμε όμω και μια ομάδα επιθεωρητών, η οποία απεστάλησαν πολλές φορές αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη που είχαν πληγεί από την ασθένεια, όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε ότι θα είχαμε σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων εξάλληψης, αλλά για να γίνονται και οι σωστοί έλεγχοι στα σύνορα, ιδίως όσον αφορά τους επιβάτες που ερχόντουσαν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλαμε εκεί πολύ αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να μην έχουμε μολυσμένα προϊόντα και υλικά, τα οποία μεταφέρουν ενδεχομένω κάποιοι πολίτες. Επίσης, χρησιμοποίησαμε εμπειρογνώμονες όσον αφορά την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, οι οποίοι πήγαν επί τόπου και δώσαν απαραίτητες συμβουλές στις εθνικές αρχές για την εξάλληψη της νόσου. Προβλέπονται όμως και προγράμματα κατάρτισης, προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις κτηνιατρικές εθνικές αρχές για να αντιμετωπίσουν και να εξαλείψουν την νόσο σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχουμε βέβαια και την παροχή επιστημονικών συμβουλών μέσω της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής με την Ασφάλεια Τροφίμων η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων και αυτή την εβδομάδα μάλιστα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα τη εμφάνιση τη νόσου στα αγριογούρουνα. Επίση συνεργαζόμαστε με το Διεθνέ Γραφείο Επιζωτιών καθώ επίση και με τη ΦΑΟ και από κοινού οι δύο αυτοί οργανισμοί έχουν δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για, την, για τον προδευτικό έλεγχο τη διασυνοριακή εμφάνιση τη ασθένεια. Συνεργαζόμαστε λοιπόν στα πλαίσια του φόρουμ αυτού και με αρχές από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Έχουν γίνει επιθεωρήσεις λοιπόν σε 7 συνολικά πλέον χώρες και στα πλαίσια των επιθεωρήσεων αυτών προσπαθούμε να δούμε ποια τακτική, ποια προσέγγιση ακολουθεί κάθε χώρα ξεχωριστά για την εξάλληψη της νόσου. Τώρα πώς έχει η κατάσταση επί του παρόντος. Έχουμε μία περιφερειοποίηση της νόσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με την εμφάνιση άλλων ασθενειών, όπως για παράδειγμα η γρήπη. Προσπαθούμε δηλαδή να οριοθετήσουμε γεωγραφικά την περιοχή αυτή, η οποία θεωρείται ότι έχει θυγεί, ότι δεν είναι απαλλαγμένη από την ασθένεια. Αυτή ακριβώς λοιπόν την περιοχή βλέπετε στην διαφάνεια αυτή και προσπαθούμε να περιχαρακώσουμε την μολυσμένη αυτή περιοχή και να την διαιρέσουμε σε τρεις επιμέρους περιοχές με κόκκινο βλέπετε τις περιοχές εκείνες όπου έχουμε κρούσματα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε αγριογούρουνα, έχουμε τη ροζ, τις ροζ περιοχές, όπου έχουμε μόνο κρούσματα σε αγριογούρουνα και έχουμε έπειτα τις μπλε περιοχές, όπου έχουμε ουσιαστικά μια ζώνη προστασίας, ένα buffer zone περιοχές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύεται από την όσο ε, προστατεύονται οι υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια διαβάθμιση και στους περιορισμούς που χρησιμοποιούμε. Πιο αυστηροί περιορισμοί στις κόκκινες περιοχές, λιγότερο αυστηροί στις ροζ περιοχές. Σε κάθε περίπτωση πάντως μέλημά μας είναι να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τις υπόλοιπες περιοχές και να μπορούμε να έχουμε εισαγωγές κρέατος ή ζών των ζώων από τρίτες χώρες ή άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν πληγεί ε, από την νόσο. Βλέπετε εδώ πέρα χρηματοδότηση περαιτέρω μέσων έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια και θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα επόμενα χρόνια. Τώρα, τόπου, όπως σας είπα, έχουν πάει οι ομάδες επιθεωρητών μας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ε, προτείνει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο βιοπροφύλαξη σε διάφορε γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Αυτό ακριβώ θέλουμε να αποφύγουμε. Να έχουμε δηλαδή κρούσματα και στίε σε συγκεκριμένε γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Ξέρετε ότι μπορούμε να έχουμε άλλες περιοχές οι οποίες είναι μολυσμένες από την νόσο, αλλά μπορεί να μην είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να οριοθετήσουμε τις περιοχές αυτές που είχε εμφανιστεί νόσος και θέλουμε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε κάποιες περιοχές απαλλαγμένες από την νόσο αυτή. Αναφέρθηκα επίσης στη συνεργασία αυτή που έχουμε ανάμεσα στο Εθνικό Γραφείο Επιζωτιών και τη ΦΑΟ έχουν λάβει χώρα ε, συνεδριάσεις στο Μίνσκ και στη Λετωνία με τις 7 χώρες που έχουν θυγεί από την Όσο, όπου είχαμε δηλαδή τους επικεφαλείς των κτηνιατρικών υπηρεσιών των 7 αυτών χωρών και προσπαθούμε ουσιαστικά να πείσουμε πλέον τη Λευκορωσία να μας δώσει πιο διαφανή στοιχεία. Ένα σημαντικό κριτήριο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει υπόψη μας είναι η χρησιμοποίηση υπολοιμάτων τροφίμων προκειμένου να τραφούν κάποιοι χείδη σε συγκεκριμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούνται πολλά υπολείμματα φαγητών πολλέ φορέ σε κάποιε γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Μέσα σε αυτά τα υπολείμματα φαγητών έχουμε μολυσμένο κρέα, το οποίο κατά αυτόν τον τρόπο μεταδίδει την νόσο σε κάποιου υγιεί κατά τα άλλα χείρου. Προφανώ η πρακτική αυτή του swill feeding, τη χρησιμοποίηση υπολείμματων φαγητών, απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε τέτοια πρακτική σε οποιαδήποτε γεωργική εκμετάλλευση. Επίσης, θέλουμε σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε να υπάρχει μία ανεξέλεγκτη απόρριψη σφαγίων ή απόθεση νεκρών ζώων, ιδίως όταν τα ζώα αυτά έχουν εμολυνθεί. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πολλές φορές τα σφάγια αυτά ψύχονται και παγώνουν, αλλά είναι σε θέση να μεταδώσουν την όσο όταν αυξάνεται η θερμοκρασία την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ε, διαχείριση των μετακινήσεων των άγριων χείρων. Ξέρετε ότι η τακτική που ακολούθησε η Λευκορωσία όσον αφορά τους, τα αγριογούρουνα το γεγονός δηλαδή ότι θανάτωναν τα αγριογούρουνα προκειμένου να αναχαιτήσουν την εξάπλωση της νόσου, αυτό είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί υπήρχαν τεράστιοι πληθυσμοί αγριογούρων που μετακινήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας και κατά αυτόν τον τρόπο μολύθηκαν τελικά πάρα πολλές περιοχές στη Λευκορωσία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για τη διαχείριση των πληθυσμών αγριογούρουνων και για αυτό το λόγο η ΕΦΣ ανέλαβε εδώ πέρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα αναφερθώ σε αυτές σε λίγο. Όσον αφορά τώρα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όταν είχαμε το πρώτο κρούσμο στη Λιθουανία στις αρχές του 2014, η Ρωσία κατευθείαν απαγόρευσε οποιαδήποτε εξαγωγή χείρων ή χείριου κρέατος από το σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα δισεκατομμύρια ευρώ αναπερίπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απλώς και μόνο η εμφάνιση του κρούσματος αυτού στα σύνορα α, Ρωσίας και Λιθουανίας ήταν ε, αρκετό προκειμένου η Ρωσία να προχωρήσει σε μια γενική απαγόρευση των ε, εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ήταν σωστή η αντιμετώπιση αυτή της Ρωσίας, ότι ήταν εντελώ δυσανάλογη και γι' αυτό το λόγο στα πλαίσια πλέον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στη Γενέβη όσον αφορά αυτά τα υγειονομικά και φυτογειονομικά μέτρα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία. Επιστημονικά στοιχεία ότι μεταξύ του πληθυσμού αγριόχειρων εξαπλώνεται η νόσος και αυτό δείχνουν τα περισσότερα στοιχεία και εκεί πρέπει να στραφούμε για την καταπολέμηση αφρικανικής πανόλης των χείρων. Ε, όχι διασυνοριακά, γιατί ε, μπορούμε να οδηγήσουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Και το έχουμε ξεκαθαρίσει και στα κρατημέλη ευθύς εξ αρχής, όσα ε, ε έχουν κρούσματα δηλαδή. Δεν είναι εύκολο όμως ένας υπουργός ε, δύσκολα μπορεί να πει μην κάνετε τίποτα, μη θανατώνετε αγριόχειρους και ε, είχαμε αυτή τη συνάντηση ο Βίλνιος με τους τέσσερις υπουργούς ε, την προηγούμενη εβδομάδα και τους περάσαμε ξεκάθαρα το μήνυμα. Οι κτηνίατροι ε, χρειάζονται επιτόπου και οι περιβαλλοντικές αρχές, ε, οι δασοφύλακες πρέπει να καταλάβουν τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρχει μεταφορά, μετακίνηση αγρόφερων από το ένα μέρος στο άλλο. Υπάρχουν διάφορες ε, στρατηγικές όπως είπα ε, που δεν είναι εφικτές και η μία ε, αναφέρθηκε ήδη θανάτωση μεγάλο αριθμό αγριόχειρων. Είναι σαν να λέμε για να αποφύγουμε τη γρήπη των πτηνών να θανατώσουμε όλα τα πτηνά. Κάτι αντίστοιχο είναι. Δεν είναι δυνατό αυτό ούτε για τα αγρία πτηνά ούτε για, τα, για τους άγριους χείρους. Άρα Μπορούμε να έχουμε στοχευμένη θύρα θηλυκών για να πέσει ο πληθυσμό και να μην υπάρχει μετακίνηση. Γιατί αν μετακινούνται μεταφέρουν ε, την νόσο. Και αν φτάσουμε σε κάποιο κατόφλιο ε, πεθαίνει από μόνη της η νόσος, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί οι ε, προσβληθέντες χείροι πεθαίνουν και δεν υπάρχει εμβόλιο. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχαμε τη δυνατότητα ε, να εκριζώσουμε νόσους ε, με τον εμβολιασμό. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει εμβόλιο διαθέσιμο και με βάση τους ε, επιστήμονες δεν υπάρχει και ελπίδα να βρεθεί στο άμεσο μέλλον ένα εμβόλιο. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα. Όπως είπα, κυνήγι, πολύ επιλεκτικό κυνήγι, αποφεύγοντας τη μετακίνηση των αγριόχειρων, απαγόρευση των ζωοτροφών, ιδίω με υπολείμματα τροφίμων. Να μην χρησιμοποιούνται δηλαδή τέτοιου είδου ζωοτροφέ σε μικρά αγροκτήματα, η απομάκρυνση των σφαγίων για να μην τρέφονται με αυτά αγριόχειροι, κάτι που συνηθίζουν κατά τα άλλα και ανθρώπινος παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός να αντιληφθεί την κατάσταση και ο νοτρόφος... Ε, και οι υπόλοιποι που πηγαίνουν Σαββατοκύριακο και περπατάνε στο δάσος, να αντιληφθούν αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορεί γυρίζοντας να έχουν ε, να γίνει φορείς αυτού του ιού, να μεταφέρουν πάνω σε αυτόν τον ιό. Τι κάνουμε τώρα στο προσεχές μέλλον. Θα αναθεωρήσουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία σας παρέθεσα πριν. Θα δούμε ε, ποια είναι η πιο πρόσφατη συμβουλή από την ΕΦΣΑ για να φτιάξουμε τη στρατηγική μας, τη στρατηγική εξόδου για την άρση των περιορισμών. Γιατί όταν ε, εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα, εξαλείφεται μεταξύ των πληθυσμών αγροχείων από μόνη τη η αλλά θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να επιτηρούμε την κατάσταση, να ενισχύσουμε την επιτήρηση και να επιβάλλουμε τη βιοασφάλεια στα αγροκτήματα. Ευχαριστώ και είμαστε στη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρος. Έχω τώρα κατάλογο με εγγεγραμμένους. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που περιλάβατε το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξή μας. Ευχαριστώ και τους ε, συντονιστές που συμφώνησαν να περιληφθεί το θέμα αυτό της Αφρικανικής Πανόλου των Χείρων που είναι τεράστια σημασίας. Δεν αρκεί να παρακολουθήσουμε μόνο την παρουσίαση του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην λάβουμε άλλα μέτρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια, την παρακολούθηση, monitoring που δεν αρκεί όμως. Χρειαζόμαστε ανάληψη δράση Και εννοώ και οι χώρε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι πιθανώ το μόνο μέλος της Επιτροπής Γεωργία που κατοικεί μόνιμα μέσα σε αυτή την ερυθρά ζώνη που δείξατε. 20 χιλιόμετρα από τον τόπο όπου διαμένω έχει ξεσπάσει η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων σε ένα αγρόκτημα και χρειάστηκε να σφαγούν και να ταφούν 20.000 χείρι. Σήμερα η αγροτική εκμετάλλευση δεν υφίσταται πλέον, διότι δεν ανανεώθηκε η αγέλη των χείρων που εξέτρεφε. Σε τρεις από δώδεκα κτηνοτροφικές μονάδες όπου έχει ξεσπάσει η νόσος, καταστράφηκε ολόκληρη η αγροτική εκμετάλλευση στην η κατάσταση, διότι δεν εξαφανίζεται η αγροτική εκμετάλλευση. Δεν το επιτρέπουν αυτό. Δεν σε αυτό το μέτρο. Εμείς το κάνουμε όμως στην χώρα μου, στη Λιθουανία. Ούτε τώρα στη Λιθουανία, ούτε στην Πολωνία δεν έχει μειωθεί ωστόσο η νόσος. Δύο τρίτα της περιφέρειας, της περιοχής όπου έχει ε, ξεσπάσει νόσος έχουν ληφθεί μέτρα. Δεν επιτρέπουν στους κτηνοτρόφους να εκδέχουν άνω των 100 χείρων. Σε περιοχές της είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κατεύθυνση η μονάδα. Έχουμε προβλήματα βέβαια και με τις κυρώσεις με τη Ρωσία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σταματήσουν αυτά για να μπορέσουμε να λύσουμε και τα προβλήματα του χείριου κρέατος. Μέχρι τώρα πάντως οι ελπίδες μας δεν έχουν δικαιωθεί. Αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε μια προσπάθεια δηλαδή στην ίδια την αγροτική εκμετάλλευση. Ο πληθυσμό των αγριόχειρων είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Στη Λιθουανία εντοπίσαμε 57 αγριόχειρους που έπασχαν από την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Υπάρχουν και αγριόχειροι που είναι φορείς του ιού χωρίς τελικά να πεθαίνουν από αυτόν ή χωρίς να εκδηλώνεται η ασθένεια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι αγριόχειροι κάποια στιγμή αναπτύσσουν ανοσία στην ε, Αφρικανική Πανόλη. Εξακολουθούν να είναι φορείς όμως. Άλλο πρόβλημα είναι η εξάπλωση της νόσου μέσω προϊόντων που εισάγονται από τη Λευκορωσία. Αντιμετωπίζουμε επίσης και ένα άλλο θέμα, το εξής. Δεν μας επιτρέπεται η εξαγωγή ζωντανών ζώων στην Πολωνία, ακόμα και από περιοχές όπου δεν έχουν σημειωθεί κρούσματα της νόσου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να εγκύψει το θέμα, αλλά ο χρόνος περνά και νέα δεν έχουμε. Ειδήσει δεν έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όχι επειδή λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις οι αρχές αλλά επειδή οι εισαγωγείς θεωρούν ότι ακόμα και με εισαγωγή άσχετων προϊόντων από, σύνολο από, σύνομα, από χείριο κρέας μπορούν να μπορεί να οδηγηθούμε σε εισαγωγή της νόσου. η κυβέρνησή μας έχει επενδύσει πολύ σε περιφράξεις στην περιοχή. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να προστατεύσουμε τις περιοχές που δεν έχουν προσβληθεί ακόμα. Μόνο οι περιφράξεις μπορούν να αποδώσουν. Αν δεν υπήρχαν οι περιφράξεις, μέχρι και η Γαλλία και το Βέλγιο και στην Γαλλία και στο Βέλγιο θα είχαν φτάσει οι μολυσμένοι χείροι. Οι μολυσμένοι αγριόχειροι δηλαδή. Βεβαίω είναι βαρύτατες οι οικονομικές επιπτώσεις. Μέχρι 75% των μέτρων αντισταθμίζονται, όχι όμως όλα. Για παράδειγμα, οι κυνηγοί αντιμετωπίζουν και αυτοί τις επιπτώσεις. Υφίστανται και αυτοί ζημίες για τι οποίε δεν αποζημιώνονται Άρα πρέπει να προβληματιστούμε, να αναλάβουμε δράση, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το οποίο μέχρι τώρα μεγαλώνει, δεν μικραίνει. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθίσει να δουλέψει πιο σοβαρά. Αν δεν αρκούν αυτά, τότε να προχωρήσουμε και στη λήψη άλλων μέτρων, γιατί μέσα στα χρόνια η γνώση εξαπλώνεται. Ο κ. Σάγνιου Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για το briefing που έκανε για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, για, το, για την οποία λέει ότι δεν υπάρχει και εμβόλιο. Ευχαριστώ βέβαια και τον Λιθουανό συνάδελφο που έχει εμπειρία από πρώτο χέρι της νόσου και που εξηγεί ένα σενάριο που μπορεί όντω να συμβεί. Λέει λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη κτηνοτροφική, χειροτροφική μονάδα έκλεισε, προκλήθηκε μεγάλη ανεργία. Εγώ στην θέση του χειροτρόφου αυτού θα έψαχνα να βρω αλλού δουλειά και μπορεί να πήγαινα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι νοητό αυτό. Το, νοητό ε, το... Ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε εξάπλωση της νόσου. Μπορεί δηλαδή να φτάσει η ε, νόσος αυτή να μεταδοθεί στο Ενωμένο Βασίλειο επειδή κάποιος ο οποίος δούλευε στη Λιθουανία και έχει μολυνθεί πηγαίνει να δουλέψει στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Εάν πρόκειται λοιπόν να φύγουν να μεταναστεύσουν το, το εργατικό του προσωπικό μπορεί να υπάρξει σημαντικός κίνδυνος. Αν φέρουν την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στην Μεγάλη Βρετανία, τότε θα κλείσει η χειροτροφική μονάδα στην οποία θα πανεργαστούν. Άρα έχουν κάθε συμφέρον οι ίδιοι να φροντίσουν ένα απόλυτα καθαρή. Αυτό που θέλω επίσης να κάνω είναι να απευθύνω μήνυμα και ε, στους υπουργούς, τους άλλους υπουργούς, διότι οι τουρίστες που πηγαίνουν να περπατήσουν στα δάση αυτή της όμορφης περιοχής της Λιθουανίας μπορεί να επιστρέψουν και να μεταφέρουν τον ιό. Μαζί λοιπόν με τα ε, ε, πραγματικά με τα ε, γνήσια συλληπιτήρια που απευθύνω στους φίλους της Λιθουανίας απευθύνω και αυτή την προειδοποίηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν ε, οικονομικές επιπτώσεις, πολύ μεγάλης κλίμακος μάλιστα, διότι αν εξαπλωθεί περισσότερο η νόσος αυτή, τότε νομίζω ότι ε, θα απειληθούν πάρα πολλές κοινοτροφικές μονάδες. Θα μπορούσαν να απειληθούν μονάδες ακόμα και στην ε, Δανία, στις κάτω χώρες. Και δυστυχώς, κανείς δεν μας είπε πώς πήγε η ασθένεια αυτή, πώς μεταφέρθηκε από τη Μοζαμβίκη στην Ευρώπη. Κέριο το ερώτημα αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι αγριόχειρος αυτός ο οποίος πήρε το πλοίο και ήρθε μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ιδίω όσον αφορά τα τρόφιμα τα οποία φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες στις οποίες αγνοούμε αν έχει εμφανιστεί μια τέτοια πανδημία. Και ξέρετε ότι υπάρχουν και χώρες όπου δεν υπάρχουν επίσημες κτηνιατρικές αρχές. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Οι χώρες αυτές δεν μας δίνουν κανένα αξιόπιστο στοιχείο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή επικρίνουμε τη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε αν και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προασπίσουμε τον δικό μας το κοινοτροφικό τομέα και να θέσω τώρα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τουλάχιστον κάπως τις αγέλες αυτές οι οποίες νόσησαν και ιδίως όσον αφορά τους χείρους. Υπάρχουν ε, δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή αποδεικνύουν ότι όντως βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, ότι όντως ακολουθούμε τη σωστή πολιτική. Νομίζω ότι η διαδικασία που ακολουθείται αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ιδιαίτερα χρονοβόρα και αναφέρομαι στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Είμαστε η τελευταία χώρα η οποία χρειάστηκε να εξαλείψει την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων και εγώ μάλιστα είχα εμπλακεί στι τελευταίε προσπάθειε που γίνανε στην χώρα μου, την Πορτογαλία, για την εκρίζωση τη νόσου αυτή. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή και ιδιαίτερα χρονοβόρα και όσον αφορά τον εμβολιασμό. Ας συνειδητοποιήσουμε το εξή. Καθότι η ασθένεια αυτή μπορεί να λάβει τεράστιες διαστάσεις, ενδεχομένως να πρέπει να αναπτυχθεί και ένα εμβόλιο για την Αφρικανική πανόλη των χείρων. Έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε την κλασική πανόλη των χείρων. Αν καταφέρναμε να κάνουμε κάτι τέτοιο μέσω ενό εμβολίου και για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, θα μειώναμε πάρα πολύ το κόστο, το οικονομικό αντίκτυπο τη ασθένεια αυτή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πέρα από την αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή εμφανιστεί η νόσος, να έχουμε και την απαραίτητη πρόληψη. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να εξαλείφουμε την νόσο αυτή. Αν είχαμε λοιπόν ένα εμβόλιο, κατά της αφρικανικής πανόλης των χείρων, θα ήταν λάθος να συνεχίσουμε την πολιτική της εκρίζωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εφιστάμενες μεθόδους και αν αναπτυχθεί εμβόλου προφανώς θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια μέτρα χρησιμοποιήθηκαν και αν χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των μέτρων των διαθέσιμων για να διασφαλίσουμε ότι ούτε ένα κιλό κρέας δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει από μολυσμένη χώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα, ποιους φραγμούς έχετε δημιουργήσει εσείς για να μην εξαπλωθεί η νόσος, τι μορφή μπορεί να πάρει αυτή η περίφραξη στην οποία αναφερθήκατε. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι εκαθάρισης μπορούμε για παράδειγμα να διασφαλίσουμε ότι συγκεκριμένε κόκκινες περιοχές ή μολυσμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, οποιοδήποτε όχημα για παράδειγμα ή άνθρωπος ή ζώο περνάει από τέτοιες περιοχές όντως απολυμμένεται. Νομίζω ότι θα πρέπει για τα οχήματα να απολυμμένονται τα λάστικα, για τους πολίτες θα πρέπει να απολυμμένονται τα παπούτσια τους, να δημιουργήσουμε δηλαδή ειδικού τάπητες απολύμανσης, πρέπει να υπάρχουν πραγματικά τέτοια μέτρα, γιατί ξέρετε ότι τελικά η νόσος μεταδίδεται πολύ περισσότερο από μικρές οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες. Εκεί θα πρέπει να επέμβουν οι υγειονομικές αρχές, εκεί θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα προφύλαξης και απολύμανσης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε διατροφική αλυσίδα μολυσμένο κρέας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο τώρα πάλι στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο επόμενο ομιλητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που εγγράψατε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι μια νόσος που αποτελεί πρόβλημα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για τις χώρες της Βαλτικής και υπάρχει και υψηλός κίνδυνος μετάδοση. Η προέλευση της ε, επιδημίας πριν από 1,5 ε, χρόνο ήταν η Ρωσία, αυτή ήταν η χώρα προέλευση. Το γεγονός ότι η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων ε, έχει εξαπλωθεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει έχει οδηγήσει και στο εμπάργκο και στο μποϊκοτάρισμα των εισαγωγών από τη Ρωσία είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε αν εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για την εκρίζωση της νόσου. Εδώ και μισή χρόνο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζει την έρευνα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά και τη μετάδοση, την εξάπλωση και τον τρόπο εκρίζωσής της. Επόμενος ομιλητής, ε, κύριος Ξυλίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είπατε, ε, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην παρουσίαση, ότι το 2007 ή στη, στη Γεωργία, είπατε, 2015 είμαστε τώρα και πολλά κράτη ε, εξακολουθούν να πλήττονται από την όσο μετά από 8 χρόνια επομένως δεν έχει ακόμη κρυζωθεί η νόσος, το αντίθετο μάλιστα, παίρνει τα πάνω της αν μπορώ να το πω έτσι. Και επειδή και η Πολωνία είναι μια από τις χώρες που πλήττεται, θέλω να αναφέρω δύο προβλήματα. Το πρώτο, ε, επειδή μιλήσαμε για τρεις ζώνες ε, και για τις υποχρεώσεις ε, των κτηνοτρόφων, για τη διάθεση των σφαγίων και για τη βιοασφάλεια αυτό τι σημαίνει, πολύ απλά ακόμη μεγαλύτερο κόστος παραγωγής ε, με τις όρους αυτούς που ε, προτείνεται τώρα και επομένως δεν είναι αποδοτικό. Δεύτερον, ε, η αντίδραση των υπηρεσιών μεταποίησης κρέατος στην Πολωνία μεγάλο μέρος είναι επιχειρήσεις με ξένο κεφάλαιο που δημοσία λένε πολύ απλά ότι δεν πρόκειται να επεξεργαστούν κρέας το οποίο έρχεται από την Πολωνία. Και δεν μιλάμε για τη μία και μόνη περιφέρεια που εντοπίστηκε το πρόβλημα, αλλά από όλη την ε, Πολωνία, από όλη την επικράτεια της χώρας. Και αυτό σημαίνει ότι και ε, μειώθηκαν πολύ σημαντικά οι τιμές του χείρου κρέατος στην Πολωνία. Ακόμα πιο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα λοιπόν δημιουργείται για τη χώρα. Με ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντέν τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευρύτερα, το ζήτημα αυτό δημιουργεί και ένα άλλο θέμα ε, της διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Ε, ε, από τη μία δηλαδή έχουμε τα δέσποτα ή τα άγρια ζώα και αφετέρου τα κατοικίδια, τα οικόσιτα. Υπάρχουν προβλήματα. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει έρευνες που μπορεί να γίνονται και θα ήθελα να επιστήσω και την προσοχή της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ στις απόψεις της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τα οικοσυστήματα. Για κάποια είδη που χθε έπρεπε να προστατευτούν σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δημιουργείται πρόβλημα της ε, διασταυρωμένη αυτή επιμόλυνσης. Εγώ έχω μια περίπτωση μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας για ένα προστατευόμενο είδο από τις Άλπεις. Η βρουκέλωση όμως ε, μεταβοηδή μεταδο, μεταδόθηκε σε αυτό το είδο και σήμερα είχαμε ε, σε παιδιά, σε δύο παιδιά κρούσματα υψηλού περαιτού που πολλοί ε, επιστήμονες πιστεύουν ότι μεταδόθηκε από τα περιτώματα ε, μολυσμένων ζώων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι η Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα ε, για τους κινδύνους διασταύρωσης, διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των οικόστων και των άγριων ζώων. Πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε ότι ε, έχουμε από τις ανατολικές χώρες ε, παράνομες εισαγωγές ε, αγριόχειρων, αγριογούρνων που είναι και γνωστό. Άλλωστε στην περιοχή δεν ξέρω αν ευθύνεται και την κατάρριξη των συνόρων. Αφού δεν υπάρχουν σύνορα ε, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριο Πέτεμαν. Χρειάζεται αντίδραση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ενία αγορά ή όχι. Ακούμε συχνά να μιλούν οι παραγωγοί για φαινόμενα στην ενία αγορά. Αλλά α, μετά λένε ενία αγορά δεν επιτρέπεται να παρέμβει κανείς. Όμως όταν πρόκειται για αφρικανική πανόλη των χείρων, τότε α, λέμε αυτό αφορά μόνο τις συγκεκριμένες χώρες, είτε είναι η Πολωνία, μετα λενε ενή αγορα δεν επιτρεπεται να παρεμβει κανεις ομως οταν προκειται για αφρικανικη πανολη των χειρων τοτε α λεμε αυτο αφορα μονο τις συγκεκριμενες χωρες ειτε την πολωνια την λιθουανια κλπ. Εφόσον έχουμε όμως ενιαία αγορά και εφόσον εμφανίζεται η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στην ε, Πολωνία, τότε αυτό αφορά και την Πορτογαλία. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει με επαρκή τρόπο. Ο κίνδυνος εμφανίζεται στην Πολωνία, αλλά εκεί αφήνουν τους ε, χειροτρόφους στη μοίρα τους δόθηκε ένα εκατομμύριο ευρώ για κάποια πρώτα μέτρα, αλλά δεν δόθηκε ποτέ επαρκής υποστήριξη. Ούτε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η Ρωσία επέβαλε αυτή την παράλογη απαγόρευση εισαγωγών, παρόλο που η νόσος ήλθε από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι αντίστροφα βεβαίω. Θέσπισαν λοιπόν αυτή την απαγόρευση εισαγωγών και δεν υπήρξε σχεδόν καμία αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα πρόκειται για πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Η νόσος θα επεκταθεί. Ήδη έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στην χειροτροφία στην Πολωνία. Μέχρι πρόσφατα η Πολωνία είχε πλεόνασμα στις εξαγωγές μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τόνους του χείριου κρέατος, τώρα έχουν φτάσει σε έλλειψη, σε έλλειμμα Πρέπει να αποζημιώσουμε τους χειροτρόφους σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από αυτό που γίνεται ήδη. Και κάτι για τον κύριο Άγνιου που ανησυχεί για τους Πολωνούς μετανάστες που θα πάνε να δουλέψουν στη Μεγάλη Βρετανία. Οι χειροτρόφοι δεν πάνε, δεν κάνουν τουρισμό στη Μεγάλη Βρετανία κύριε Άγνιου, μην ανησυχείτε. Bardzo proszę pan poseł Agniu, ο πρόεδρος. Κύριε Άγνιου, ναι, αφού ακούσατε το όνομά σας. Ναι, ναι, δεν μιλούσα για Πολωνούς τουρίστες που θα πάνε στην ε, ε, Μεγάλη Βρετανία. Είπα ότι ενδέχεται απολυμένοι εργάτες χειροτροφίων στην Πολωνία μπορεί να σηκωθούν να πάνε να βρουν δουλειά στο Ενωμένο Βασίλειο ή το ίδιο οι Λιθωνοί και να μεταφέρουν τον ιό. Μήπως δεν μεταφραστές, λέει ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ, Χόισλινγκ. Τι θα κάνουμε, νέου φραγμού στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουμε την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Δεν μου φαίνεται το μέτρο αυτό να είναι πιστικό. Τα όσα προτείνει πάντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε και αυτά μου φαίνονται πολύ πιστικά. Διότι από την τελευταία συζήτηση η περιοχή εξάπλωση της νόσου έχει μεγαλώσει. Άρα τα μέτρα είναι όντω επαρκή. Ούτε με επίθετε πολύ με αυτά με τους αγριόχειρους. Να απαντήσετε σε αυτά που είπε ο κ. Κρουπέ. Αναπτύσσουν ανοσία οι αγριόχειροι στον ιό. Και τι γίνεται. Ψοφάνε εφόσον έχουν μολυνθεί. Αν γίνονται, αν αποκτούν ανοσία, τότε την άλλη υπόθεση. Εκεί γίνεται τελείω διαφορετική συζήτηση. Γιατί άραγε είναι αδύνατον να βρεθεί κάποιο εμβόλιο. Φταίει το ότι οικονομικά δεν είναι ενδιαφέρον για την ε, φαρμακοβιομηχανία. Τεχνικά δεν πιστεύω να είναι το πρόβλημα. Τεχνικό δηλαδή δεν πιστεύω να είναι το πρόβλημα. Χρειάζεται ίσως κάποια υποστήριξη για την ανάπτυξη του εμβολίου. Και μια παράκληση. Χρειάζεται μεγαλύτερη, περισσότερη ενίσχυση Τη αγροτική οικονομία στι περιοχέ αυτέ. Δεν είναι δυνατόν τώρα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ούτω ή άλλω πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο, να ε, υφίστανται και τι επιπτώσει τη ε, ζωνό αυτή. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια στην περιοχή αυτή. Σα ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση, λέει ο πρόεδρο. Πώ αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κίνδυνο μόλυνσης. Εδώ η νόσος υπερβαίνει κάποια βιολογικά όρια, σύνορα αν θέλετε. Έχετε το λόγο. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις που καλύπτουν και όλο το φάσμα της ε, παρουσίασης που έκανα. Ας αρχίσουμε από την αρχή από τη Μοζαμβίκη ξεκίνησε η νόσος, ναι. Έφτασε στη Γεωργία από τα κατάλοιπα της κουζίνας, της ε, παρασκευής τροφίμων δηλαδή, στην κουζίνα ενός πλοίου που ερχόταν από τη Μοζαμβίκη και όπου δεν κατεστράφησαν αυτά. Υπάρχουν, ε, αυστηροί, υπάρχουν αυστηρές απαγορεύσεις για τα υπολείμματα τροφών που φτάνουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλοία ή από αεροσκάφη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καταστραφούν. Το ίδιο ισχύει και για προσωπικές εισαγωγές κρέατος από, την... από περιοχές. Δεν μπορείτε καν να φέρετε ένα σάντουιτς τέλος πάντων μέσα ε, ε, ε, από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι στα προϊόντα αυτά μπορούν να κρύβονται νόση υπενθυμίζω ότι και η μεγάλη ε, ε, επιζωτία στο Ενωμένο Βασίλειο του Αυθόδου πυρετού στο Ενωμένο Βασίλειο προήλθε από παράνομο swill feeding κοντά στο Κάσλ. Swill, δηλαδή υπολείμματα τροφών που προήλθαν από την κουζίνα ενός πλοίου που δεν, από το μαγειρίο ενός πλοίου που δεν καταστράφηκαν. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνο, Εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος. Γι' αυτό και έχουμε τόσο αυστηρούς κανονισμούς είτε για νόμιμε, εισαγωγέ, είτε για όσα μεταφέρουν οι επιβάτες πλοίων κλπ. Εν προκειμένου θέλω να τονίσω ακόμη ότι το χοιρινό κρέας επιτρέπεται να εισάγεται να εισάγεται στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο από 8 τρίτες χώρες ανά τον κόσμο. Άρα, παράνομες δραστηριότητες οι οποίες παραμένουν παράνομες. Εδώ όμως παίζει ένα ρόλο και η άγρια πανίδα. Έχουμε και την πύρα της ε, γρήπης των πουλερικών που μεταδόθηκε καθώς και του ιού ΙΤΑ7N7 στο Ενωμένο Βασίλειο πάλι, ο οποίος ε, οδήγησε στην καταστροφή μεγάλου αριθμού πουλερικών στην Μεγάλη Βρετανία. Άρα τα άγρια ζώα εμφανίζουν τον κίνδυνο αυτό. Αλλιώ υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι βεβαίω. Αναφέρθηκε μια μεγάλη χειροτροφική μονάδα στη Λιθουανία. Όντω, για μας είναι μυστήριο. Η βιοασφάλεια ήταν σε υψηλό επίπεδο στην μονάδα αυτή. Στείλαμε και αποστολή προ 10 ημέρου και γνωρίζουμε πόσο ισχυρός, πόσο δυναμικός είναι ο ιός αυτός και στην φύση. Μπορούν να φτάσει, μπορεί να φτάσει ο ιός και στις ε, ε, μπότες των διαφόρων που κινούνται στο δάσος και ακόμα και μετά από ε, καθαρισμό τους να φτάσει στην ε, μονάδα. Άνθρωποι οι οποίοι πάνε στο δάσος μπορούν να φέρουν στα υποδήματά τους μετά τον ιό. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε δαπανίσει 4 εκατομμύρια ευρώ για αύξηση του επίπεδου ευαισθητοποίησης όχι μόνο των κτηνοτρόφων, των γεωπόνων, αλλά και των απλών πολιτών που πηγαίνουν ένα περίπατο στο δάσος στο Σαββατοκύριακο. Προσωπικές εισαγωγές. Άλλο θέμα αυτό. Ορισμένοι εξημών αναφερθήκατε σε πρόσωπα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέροντας ένα σάντουιτς. Αυτό είναι παράνομο. Δεν επιτρέπεται να το πράττουν και για το σκοπό αυτό έχουμε ζητήσει επίσης από τις χώρες μέλη να αυξήσουν την επαγρύπνηση στα σημεία διαβάσεως των συνόρων και να ευαισθητοποιούν τον κόσμο, να γνωστοποιούν στο κοινό ότι δεν επιτρέπεται να εισέρχεται με τρόφιμα. Είναι πολύ σοβαρή η νόσος αυτή και εδώ το κλειδί για να αντιμετωπιστεί είναι η biosecurity. Ερώτημα τώρα, εάν κάνουμε αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά αυτά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε για πολύ περισσότερα. Περισσότερες επιθορήσεις, περισσότερες επιστημονικές συμβουλές από ό,τι έχουμε κάνει σε οποιαδήποτε άλλη επιζωοτία. Οι επιθεωρητές μας έχουν πάει επί τόπου πάνω από 15 φορές. Εμπειρογνώμονες του ΦΑΟ και του OIE έχουν επισκεφθεί επίσης τις περιοχές που έχουν προσβληθεί. Υπάρχει και πρόγραμμα εκπαιδευτικό. Έχουν οργανωθεί μεγάλες εκδηλώσεις στις τέσσερις πληγήσεις χώρες και η ΕΦΣΑ επίσης, European Food Safety Authority, δουλεύει non-stop για το θέμα αυτό και έχουν δημοσιεύουν μάλλον σύντομα και άλλη έκθεση σύμβουλων για να οργανώσουν καλύτερα την ανταπόκρισή μας στον κίνδυνο αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ζώνες, είπα ότι μετά το καλοκαίρι θα επανεξετάσουμε την κατανομή σε ζώνες που έχουμε κάνει ως τώρα. Αναμένουμε να κορυφωθεί η εξάπλωση της νόσου το καλοκαίρι, όταν τα νεαρά άγρια χειρίδια θα εγκαταλείψουν πλέον την αγέλη και θα ε, κοιτάξουν να εγκατασταθούν αλλού. Αυτό ίσως είναι πηγή Εξάπλωση της νόσου. Θα περιμένουμε λοιπόν μετά το καλοκαίρι να επανεξετάσουμε τις υφιστάμενες ζώνες. Τώρα, οι περιορισμοί, οι ισχύοντες περιορισμοί, τα συζητήσαμε αυτά με τους τέσσερις υπουργού των φυγωμένων ε, χωρών στη Λιθουανία. Επιτρέπουμε μετακίνηση προϊόντων μεταξύ ζωνών που έχουν το ίδιο καθεστώς στις ε, χώρες αυτές. Προϊόντα δηλαδή από την ροζ ζώνη στην Πολωνία επιτρέπεται να πάνε στην ροζ ζώνη της Λιθουανίας και το αντίστροφο. Τώρα, το εμπάρκο των Ρώσων. Βεβαίως αυτό μας ευνηδίασε. Αντιδράσαμε όσο μπορούσαμε. Δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι δεν αντιδράσαμε στο εμπάρκο. Είπα στην διάρκεια της παρουσιάσεώς μου ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κινούμεθα με κατάθεση προσφυγής κατά άλλης χώρας, κατά τρίτης χώρας, στα πλαίσια του SPS. Και όπως είπα, αναμένουμε τα αποτελέσματα του πάνελ του ΠΟΕ αρχάς του επόμενου έτους. Τώρα, άλλο εμπάργο από τρίτη χώρα, ιδίως σχετικά με την Πολωνία, όπου διάφορες τρίτες χώρες έχουν απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων από ολόκληρη την επικράτεια της Πολωνίας. Και εκεί αγωνιζόμεθα κατά τις, ε, κατά, δηλαδή αντιδρούμε τις χώρες αυτές και στην Ιαπωνία πιο συγκεκριμένα. Ο Πολωνός υπουργό πήγε προ λίγων εβδομάδων στην Ιαπωνία για να προβάλλει τα σχετικά επιχειρήματα. Άρα, έχουμε και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν δεχτεί τα επιχειρήματά μας. Υπάρχουν όμως και μεγάλες τρίτες χώρες οι οποίες μας εμπιστεύονται, δεν λαμβάνουν μέτρα. Για παράδειγμα, Καναδάς, Ενωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Οι χώρες αυτές δεν έχουν λάβει μέτρα κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, γνωρίζοντας καλά ότι η αρχή της περιφερειοποίησης εφαρμόζεται ορθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στις εξαγωγές μας. Να τονίσω εδώ ότι οι περιορισμοί που έχουμε επιβάλει στις τρεις ζώνες των διαφόρων χρωμάτων ισχύουν και για εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Δεν εξάγουμε λοιπόν προς τρίτες χώρες προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνω δε φόρο τιμή στις χώρες αυτές. Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. όπως είπα πριν που δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εισαγωγές στις χώρες αυτές ε, πολωνικών προϊόντων χειρίου κρέατος. Εμβολιασμό, Για την ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο. Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά με το εμβόλιο αυτό. Τα τελευταία 30-40 χρόνια συνεχίζεται η έρευνα αυτή. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο διατέθηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα αυτή τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι οι επιστήμονες δεν βρίσκουν αντισώματα, δεν μπορούν να εντοπίσουν αντισώματα δηλαδή που αναπτύσσονται. Έτσι λοιπόν για την ώρα δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο και όπως είπα και προηγουμένως οι επιστήμονες δεν βλέπουν για το προσεχές μέλλον τη δυνατότητα να αναπτυχθεί εμβόλιο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε χρηματοδοτικά και τις ε, χώρες που έχουν πληγεί. Τα τελευταία ε, χρόνια έχουμε διαθέσει 80 εκατομμύρια ευρώ, θα συνεχίσουμε να δίνουμε λεφτά και τα επόμενα χρόνια συμπεριλαμβανομένων μέτρων που δεν προσφέρονται συνήθως για χρηματοδότηση του κτηνιατρικού τομέα. Μίλησα και για το θέμα των άγριων χείρων δηλαδή εντοπισμός και σύλληψη των αγριόχειρων και εξέτασή τους κτλ. Αυτά θα συνεχιστούν και στο προσεχές μέλλον. Νομίζω ότι όντω κάλυψα τα περισσότερα, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι προφανώς θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε πόσο προετοιμασμένοι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε την τεράστια αυτή απειλή. Ξέρετε ότι το είπατε και εσείς μπορεί να κλιμακωθεί στο μέλλον η εμφάνιση της νόσου αυτής. Στόχος μας πολλές φορές είναι στα πλαίσια της εξάλληψης να πρέπει να θανατώσουμε πολλές φορές όχι χιλιάδες αλλά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον αλλά θα πρέπει και να καταλάβουμε καλύτερα και την κατάσταση και να την καταλάβει βέβαια και η κοινή γνώμη. Και αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Άγνιου. Η μόλυνση μπορεί να γίνει μέσω μεταφοράς, μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Και παράλληλα βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους κτηνοτρόφους, τους γεωργούς, οι οποίοι απομίζονται πολύ συχνά το κόστος της νόσου αυτής. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, κτηνοτρόφοι που έχουν πραγματικά χρεοκοπήσει εξαιτία τη νόσου αυτής. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση, προφανώ. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε στα πλαίσια της κοινή αγοράς να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα δεινά. Σα ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συναδέλφου. Ολοκληρώνουμε την συζήτηση για αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης και ολοκληρώνουμε και το δημόσιο τμήμα της συνεδρίασής μας. Περνάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Να σας υπενθυμίσω απλώς σήμερα το απόγευμα να φέρετε και τις κάρτες ψηφοφορίας, γιατί από τις 3 και μετά θα ψηφίσουμε. Ας παραμείνουν λοιπόν μόνο οι συντονιστές τώρα στην αίθουσα για τη συνεδρία των συντονιστών.